going to London tomorrow morning, so I will not be there. Will you be here for the vote? No. Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. αλλά πρέπει να ξέρουν οι βοηθοί κυρίως ότι είναι ενδεικτική απλώς η ημερήσια διάταξη. Καμιά φορά πάμε πιο γρήγορα, καμιά δε αργότερα. Ο κύριος Στάιλερ μάλιστα ζήτησε να αλλάξουμε τα θέματα 9 και 10 μεταξύ τους. Είναι εισηγήτρια και για τα δύο να αλλάξουμε τη σειρά γιατί μπορεί να χρειαστεί να φύγει νωρίτερα. Όχι να μην αλλάξουμε τη σειρά, να τα βάλουμε νωρίτερα. Σας προειδοποιώ λοιπόν, μπορεί να χρειαστεί να τα συζητήσουμε ένα τέταρτο νωρίτερα από ό,τι νομίζατε. Αλλά αυτά όλα είναι ενδεικτικά, ενδεικτικά είναι. Λοιπόν, αύριο τη αιτήση του κ. Λαπάς του Δεσιάς, μετά από την ψηφοφορία για τα καλώδια, για τα χοντρά καλώδια, θα συζητήσουμε για τα τελεφέρικα. Μήπως μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη έτσι όπως, ε, όπως κατήντησε λοιπόν. Είπαμε το 9 με το 10 θα αλλάξουν λοιπόν. On announcements, um, first of all reminding you that this is... Θέλω επίσης να σε υπενθυμίσω ότι αυτά αναμεταδίδονται ότι τα έγγραφα είναι όλα στην εφαρμογή ή τα συνεδρίαση. Ανακοινώσεις μετά από 3,5 χρόνια συνεργασίας η Τζούλια Μπέργκερ μεταφέρεται στο γραφείο του Γενικού Γραμματέως Νομίζω πολύ καλό είναι αυτό και σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε για μας ιδίως για τις δημόσιες πραμήθειες. Αφού θα παραμείνει στο κοινοβούλιο πάντως θα μπορούμε να σου θέτουμε ερωτήματα. Η Ελένα Μαντάρη επίσης έχει πάρει γονική άδεια και αντικαθίσταται προσωρινά από τον Πάμπλο. Εκεί, εκεί κουνάει το χέρι του. Εκεί, εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Μετά την αποστολή στη Λετωνία έγινε αναφορά και έκθεση που θα διατεθεί μετά τις 26 Μαρτίου σε όλες τις γλώσσες. Τώρα, από τώρα όμως υπάρχει στα αγγλικά. Τώρα για τη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών δύο ενδιαφέροντα θέματα. Ένα, έγγραφο για τους τριμερείς διαλόγους με 26 συστάσεις για το πώς να γίνονται καλύτερα. Μερικοί πρόεδροι όπως και εγώ είπαμε ότι πρέπει οι τριμερείς διάλογοι να διατηρούν κάποιο ευελιξία γιατί καμιά φορά είναι μακρύτεροι από ό,τι νομίζουμε, άλλες φορές θα έπρεπε να υπάρξει μια διακοπή για να περιμένουμε περισσότερη πληροφόρηση και αν πάψει να ισχύει αυτό νομίζω ότι θα ήταν αρνητικό. Επίσης πρέπει να έχουν τον χρόνο οι συνάδελφοι και τη δυνατότητα να συνεννοούνται με άλλους ενδιαφερόμενους um. κατά τη διάρκεια των τριμερών. Πρέπει λοιπόν να βρούμε και έναν άλλο τρόπο παρουσίασης των εγγράφων εκτός από τα, το τετράστιλο. Τελεία. Επίσης έγινε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Τίμερμανς για την καλύτερη διευθέτηση, καλύτερη νομοθεσία. Και η διάσκεψη των Προέδρων ασχολήθηκε επίσης με αυτό. Είναι σημαντικό νομίζω οι εμπειρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών να ακουστούν όπως πρέπει όχι μόνο στη διάσκεψη των Πρόεδρων. Ας πούμε ο κύριος Τίμερμανς ενδιαφέρεται να δει πώς μπορεί να γίνουν καλύτερες αξιολογήσεις τύπου κατά τη διάρκεια της εξέτασης μιας νομοθετικής πρότασης. Εμείς το κάναμε αυτό και μεταξύ δύο τριμερών διαλόγων για θέματα που μπορεί να μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και του άρεσε αυτό να γίνει δηλαδή ίσως και μια άλλη αξιολόγηση να γίνεται πριν τον τελικό αποχαιρετισμό του τριμερούς διαλόγου. Αυτά όμως θα τα πούμε με τους συντονιστάς και με τις ομάδες να δούμε πώς θα συνδυαστούμε με αυτό το όλο θέμα της καλύτερης νομοθεσίας. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μου. Εγκρίνουμε λοιπόν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Θα εγκριθούν εάν δεν ακουστούν διαμαρτυρίες μέχρι την αλήξη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Το 4 τώρα, το 4 είναι ενημέρωση για τον τριμερή διάλογο για τα ταξίδια πακέτα. Thank you very much. Thank you so much. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ο Λάγκεν δεν μπορούσε να έρθει και γι' αυτό μου ζήτησε να σας πω εγώ ότι για να προχωρήσει το θέμα προτείνονται συμβιβασμοί προς το Συμβούλιο. Μια δέσμη συμβιβασμών για τους ορισμούς των οργανωμένων ταξιδιών και την περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας. Είναι η μέθοδος click-through, όπου θα μπορεί ο ταξιδιώτης να αλλάζει ορισμένα στοιχεία από τον υπαλογιστή του. Είναι ισοτικό να γνωρίζουμε ότι ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή δεν ξέρει αν κλείνει ολόκληρο πακέτο ή τίποτα λιγότερο. Ενώ με αυτά τα click-through θα υπάρχει ίση μεταχείριση όλων ως δέσμης, ως πακέτου. Αυτό έχει μεγάλη προτεραιότητα και για τους σκιώδεις και για τον κύριο εισηγητή. Άλλο βασικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων. Η εξαίρεση των ε, ταξιδιών, των επαγγελματικών ταξιδιών από το εύρος αυτού του σχεδίου. Είναι εύκολο να καθοριστούν κριτήρια και με σαφήνεια νομική. Εφόσον επαγγελματικά ταξίδια θεωρούνται όσα βασίζονται σε, ένα, σε μια συμφωνία πλαίσιο. Δεν θα μπορέσουμε όμως να καλύψουμε όλους τους επαγγελματικώς ταξιδεύοντας και μπορεί εύκολα να υπάρξουν καταχρήσεις. Εξάλλου ένα σύστημα που θα καλύπτει και τα δικαιώματα των ταξιδιωτών αυτών δεν το έχουμε. Δυστυχώς το Συμβούλιο εδώ αποδεικνύεται πολύ άτεγκτο και ο εισηγητής αποσαφήνισε ότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει συμφωνία τον Μάιο παρά μόνο εάν το Συμβούλιο επιδείξει ανοιχτό πνεύμα προς την θέση του Κοινοβουλίου και μετατοπιστεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι τεράστια σημασίας για τον εισηγητή και γι' αυτό πρέπει τα μικρά ξενοδοχεία καθώς και τα μικρά ταξιδιωτικά πρακτορία να μην επιβαρυνθούν πάρα πολύ. Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες που κλείνονται μετά από την αρχική συμφωνία δεν πρέπει να θεωρούνται τμήμα ενός πακέτου. Η δημιουργία ενός πακέτου δεν ταυτίζεται με οποιαδήποτε ταξιδιωτική υπηρεσία που κλείνεται αργότερα. Γιατί αλλιώς τα μικρά ξενοδοχεία δεν θα μπορούν πια να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ιδίως σε περιπτώσεις πτωχεύσεων. Η συγκήτρια θεωρεί ότι θα βρεθεί λύση και ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο ώστε η Λετωνική Προεδρία να μπορέσει να υποβάλει το θέμα στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας τέλη Μαΐου. όλα αυτά, πρέπει το Συμβούλιο να επιδείξει κάποια καλή θέληση και να κάνει υποχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για μια καλή περιγραφή του τι συνέβη. Θα τα χρησιμοποιήσουμε στον τριμερή διάλογο. θα δούμε τι υπάρχει στα κράτη-μέλη και αν υπάρχουν κάποιες διαφορές θα πρέπει να γεφυρωθούν. Θα το ελέγξουμε λοιπόν αυτό και στα πλαίσια της εντολής μας σαν κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Περνάμε τώρα για την επόμενη έκθεση ε, στην οποία θα κληθούμε να ψηφίσουμε αύριο. Η Όλγα έχει το λόγο. Ομιλώ την τσεχική, λέει η κυρία Σενάλοβα. Καταρχάς μπορώ να σας ενημερώσω ότι στις 2 Μαρτίου το Συμβούλιο υιοθέτησε στην πρώτη ανάγνωση την θέση του για τα συστήματα ε, χρήσης, πρόβλεψης χρήσης ε, του αριθμού 112. Έχει προϋπάρξει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του προηγούμενου χρόνου και στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου και υπάρχει μια συμβιβαστική λύση η οποία πέρασε και από τη δική μας Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα τα κράτη-μέλη Υιοθέτησαν λοιπόν την απόφαση αυτή η οποία μας επιτρέπει να περάσουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Ο κανονισμός αυτός αποτελεί τμήμα συγκεκριμένου πακέτου για την λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής κλήσης e-call θα μπορεί να χρησιμοποιείται από όλα τα οχήματα ανεξαρτήτως τύπου και ανεξαρτήτως χώρας, προέλευσης και παρουσίας. Τα συστήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αν υπάρξει ένα σοβαρό ατύχημα η κλίση να γίνεται με αυτόματο τρόπο, με μηχανικό αν θέλετε τρόπο σεβόμενοι βέβαια τις βασικές αρχές ε, προστασίας της ιδιωτικότητας. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να δεχθούμε τις προτάσεις του Συμβουλίου χωρίς περαιτέρω αλλαγές έχω την αίσθηση γιατί ανταποκρίνονται στην εντολή και στις απόψεις μας. Το σύστημα λοιπόν θα πετύχει το στόχο του να μειώσει τους τραυματισμούς και τους θανάτους στην οδική ε, μετακίνηση. Ευχαριστώ την Προεδρία, ευχαριστώ και την προηγούμενη Προεδρία, την Ιταλική, για την επικοδομητική της τάση. Ανέσα Πολύλο. Ανέσα Πολύλο. Γεια σου Βανέσα, τι γίνεται. Ε, εξ ονόματος του Συμβουλίου σας κατευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι ανάμεσά σας για την εξέταση της θέσης του Συμβουλίου γύρω από το σύστημα e-call. Είναι πολύ σημαντικό το σύστημα αυτό και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ε, πρώτο βήμα για τη μείωση του αριθμού των θυμάτων ε, στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Μειώνει λοιπόν το κόστος ε, των ατυχημάτων, μειώνει γενικά τις αιτίες των ατυχημάτων και αποδεικνύει, εν πάση περιπτώσει, με ξεκάθαρο τρόπο την τεράστια προσπάθεια που κάνουμε ε, σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Πολύ συχνά ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης δεν γνωρίζει τις προσπάθειες που γίνονται για την καλυτέρευση της ζωής του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, όσο εξοπλίζονται τα οχήματα με το συγκεκριμένο σύστημα, νομίζω η αξία αυτής της ρύθμισης θα φανεί σε όλους τους πολίτες. Sottolinea la fruttuosa collaborazione che abbiamo avuto nel quadro del processo di codecisione. Vi è stata una chiara comprensione Νομίζω ότι ε, έχει υπάρξει κατανόηση των δισταγμών και των ανησυχιών οι, οποία, ε, οι οποίες είχαν εκφραστεί. Φροντίζουμε όμως την ανθρώπινη ζωή ε, επιταχύνοντας και τις νομοθετικές διαδικασίες. Ήταν πολύ θετικό που πήρα μέρος στην διαδικασία αυτή και ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια για την προσπάθειά της και φυσικά και την Επιτροπή σας και την Πρόεδρο. Να ευχαριστήσω λοιπόν και την Επιτροπή που διευκόλυνε τη συμφωνία και την Γραμματεία που οργάνωσε τους τριμερείς διαλόγους με ταχύτατο και αποτελεσματικό τρόπο. Thank you. And would the commission... Σας ευχαριστώ. Η Επιτροπή θα ήθελε να παρέχει το λόγο. Thank you. Σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανέλθει στα θέματα πολιτικής συμφωνίας που πέτυχε το Συμβούλιο και η Επιτροπή σας. Είναι καλή η συμφωνία και η συμβασμός. Θα πρέπει να συντονιστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το e και χάρη στη δέσμευση αυτή ξεκίνησε και ξεκινάει πλέον πραγματικά αυτή η πανευρωπαϊκή ιδέα του e Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν και να ευχαριστήσουμε και ιδιαίτερα στην κυρία Σνάλοβα. Σας ευχαριστώ. Κανένα από του κοιόδες θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ο Κάρλο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχά. να ευχαριστήσω ευχαριστώντας ε, την συνάδελφο Σνάλαβα για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Να ευχαριστήσω για τις διάφορες προεδρίες, την Ιταλική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προσπάθειες που κατέβαλαν προκειμένου να διευκολυνθεί η εργασία μας. Αν υπάρχει ένα καλό παράδειγμα συναπόφασης, συνεργασίας υπό εξαιρετικές συνθήκες με αλληλοκατανόηση και διάθεση ανοιχτή, αναμφίβολα ήταν αυτή η προκειμένη περίπτωση. Κυρία Πρόεδρε, το σύστημα E-Call ε, σώζει ζωές. Τη στιγμή που πολλοί λένε ότι δεν χρειαζόμαστε πιο πολύ Ευρώπη, η νομοθεσία για το σύστημα για την εφαρμογή και την κατάσταση των συστημάτων αυτών αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς πιο πολύ η Ευρώπη μπορεί να δώσει πιο αποτελεσματικές λύσεις σε σημαντικούς τομείς όπως είναι η μείωση των αυτοκινητιστικών και η βελτίωση των υπηρεσιών σε θύματα τροχαίων. Η συμφωνία λοιπόν αυτή αποτυπώνει το συμβιβασμό Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και μπορούμε να είμαστε περήφανοι όλοι για τους στόχους που θέσαμε, τους στόχους που έχουμε ορίσει στον τομέα της ασφάλειας της τροχέας. Το γεγονός ότι είναι υποχρεωτικό το σύστημα e-call, υποχρεωτική η χρήση του πανευρωπαϊκού αριθμού από το 2018 και μετά, θεωρώ ότι θα μεταμορφώσει το τροχαίο το οποίο και την προστασία των πολιτών. Ως εισηγήτρια, η κυρία Σενάλαβα ήδη το τόνισε και θα ήθελα και εγώ να το τονίσω ότι αυτό χρειάζεται για τις κατεπίχουσες υπηρεσίες βοήθειας ιδιωτών. Θα πρέπει να υπάρχουν διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. Δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ούτε να ανταλλάσσονται σε ιδιωτικά συστήματα. Άρα, πραγματικά πρόκειται για εξαιρετικό δείγμα συνεργασία. Ευχαριστώ. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια στις 28 Απριλίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλους σας. we're going to move straight on to, um, okay, fantastic, that's really helpful. So, um, we, we are going to move straight on to... Να περάσουμε λοιπόν κατευθείαν στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εγκαταστάσεις με σχηματόρυσκημα. Εισηγητής ο κύριος Λόπες Ιστούρις Βουέτ, Αντώνιο. Δεν είναι εδώ, αλλά το ήξερα αυτό. Μας είχε ενημερώσει τον αντικαθιστά ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Δεν αντικαθίσταται από εμέ, λέει η κυρία Χόενστάιν. Αλλά μου έστειλε ναι. μία επιστολή την οποία καλούμε να σας διαβάσω. Γιατί κάτι συνέβη την τελευταία στιγμή και δεν μπορεί να είναι παρόν. Το κείμενο που μου έστειλε λοιπόν πριν λίγα λεπτά λέει το εξής. Λυπάται ο κύριος Λόπες Ιστούρης γιατί δεν μπορεί να είναι παρόν και γι' αυτό καλούμε να σας ενημερώσω για τα εξή θέματα σχετικά με τις συμβιβαστικές τροπολογίες. 141 τροπολογίες κατατέθησαν στην πρόταση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συνάδελφοι Ίνκο καθέθεσαν θέσαν 40. Το θέμα των εγκαταστάσεων με σύρματόσχηνα είναι ένα εξειδικευμένο θέμα, ένα ιδιαίτερα τεχνικό θέμα. Ο συνάδελφος Αντώνιο είχε πάρα πολλές συναντήσεις με τους συναδέλφους που κατέθεσαν τις τροπολογίες. Όλες οι τεκμηριωμένες και τεχνικά αποδεκτές τροπολογίες ε, γίνονται δεκτές. Μόνο πολύ λίγες από τις τροφολογίες αυτές δεν θα έλεγα ταιριάζουν στην διαδικασία εναρμόνισης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και δεν υποστηρίζονται από τον Αντώνιο. Υπάρχει μία μόνο συμβιβαστική μαζί με τον συνάδελφο Ζουβά και Νταντά για τα συστήματα πέδησης των εγκαταστάσεων αυτών έτσι ώστε διαφορετικές τεχνολογίες για τα συστήματα πέδησης να συνυπάρχουν στις αγορές. Οι συνάδελφοι και οι Γάλλοι συνάδελφοι κάνουν μία πρόταση η οποία ε, κάνει δεκτή την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας και εξασφαλίζει δίκαιο ανταγωνισμό σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. Έχω εδώ και το κείμενο της συμβιβαστικής τροπολογίας να σας το διαβάσω. Στις εγκαταστάσεις σειρματοσκήνων θα υπάρχουν συστήματα πέδησης μονά ή διπλά, έτσι ώστε να μπορούν να σταματήσουν το βάρος του μηχανισμού. Θα πρέπει να συντονίζονται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αντικαθιστούν το ενεργό σύστημα αν αμφισβητηθεί η αποτελεσματικότητά του. Πρόκειται για το τελευταίο λοιπόν μέσο πέδησης το οποίο θα πρέπει να αφορά και να ενεργεί στις τροχαλίες ακόμα και στην κινητήρια μονάδα του μηχανισμού. Τέλος ο κύριος Λόπες Ιστούρης θέλει να αναφερθεί στην σωστή συνεργασία με όλους τους συναδέλφους που πήραν μέρος σε αυτήν την έκθεση η οποία θα ψηφιστεί νομίζω ομόφωνα αύριο. Νομίζω ότι τελείωσα, λέει η κυρία Χόχενστάιν. There from uh, Mr. Υπάρχουν και κάποιες άλλες παρατηρήσεις από τον κύριο Λόπες Ιστούρις White. Um, where he once again would Θέλει να σας ευχαριστήσει για την συνεργασία που επιδείξατε και να ζητήσει την υποστήριξή σας ακόμα και από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ που εκπροσωπήσατε τον κύριο Λόπες Ιστούρις White την τελευταία στιγμή Λοιπόν, σας ευχαριστώ που μεταφέρατε τα σχόλιά του. Νομίζω ότι παρακολουθεί αυτά τα οποία λέμε τώρα και έχει συνεργαστεί πράγματι στενά και με τους υπόλοιπους σκιώδες. Άντερσον. Ευχαριστώ, και τους Ευχαριστώ και του ΕΛΚ που ικανοποιήθηκαν τόσο πολύ με την δουλειά του Αντωνίου. Είναι τεχνική βέβαια η έκθεση, αλλά πολύπλοκη, πολύπλοκη. Και το θέμα της ασφαλείας των προϊόντων γενικότερα, αλλά ειδικά εδώ που είναι θέμα μεταφορών, είναι ακόμα πιο σημαντικό. Παρά το ότι είναι τεχνικό λοιπόν το θέμα, θα έλεγα ότι η ασφάλεια είναι το κυριότερο πρόβλημα. Ιδίω διότι οι επιπτώσεις ενός ατυχήματος στα τελεφερίκ μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Και στόχος μας είναι να υπάρξει μία νέα διευθέτηση στο μέλλον για αυτά. Συμφωνήσαμε για τα περισσότερα στοιχεία της εκτίμησης μέσα των τροπολογιών Υποστηρίξαμε και τη συμβιβαστική που ήταν πολύ δύσκολο θέμα και υπήρξαν και πάλι υπήρξαν διαφωνίες. Πάντως το αποτέλεσμα γενικά είναι καλό. Οι περισσότερες τροπολογίες εγκρίθηκαν και νομίζω ότι παρά το ότι είναι μέτρο εναρμόνισης από την ομάδα μου εξετάσαμε και θέματα της θέσης του Κοινοβουλίου για τα ασφάλεια των προϊόντων γενικότερα γιατί εκεί δεν υπήρξε απόλυτη ταύτιση απόψεων ως προς την ερμηνεία της ρήτρα ε, φρόνησης. Αλλά καταλήξαμε πάντως σε μια θέση αποδεκτή και νομίζω ότι είμαστε σε καλή, είμαστε σε θέση τώρα να προχωρήσουμε τον τριμερή διάλογο. Στο Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι πολύ σύντομο δεν καταθέσαμε τροπολογίε. Υποστηρίζουμε γενικότερα τη συμβιβαστική τροπολογία και τη θέση της συγκητή. Βέβαια με μερικές από τις τροπολογίες, καμιά δύο μπορεί να έχουμε προβλήματα, αλλά θα τις καταψηφίσουμε δεόντως χωρίς άλλα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι. Να το πείτε παρακαλώ, να το μεταφέρετε. Και υποστηρίζουμε και εμείς τη συμβιβαστική για τα breaking systems, για τα παιδι, συστήματα παιδισης. Και ελπίζουμε ότι η συνεργασία που σημειώθηκε σε αυτή τη συζήτηση θα γίνει τελικά κανόνας. Πέρα από τη συμβαστική τροπολογία νομίζω ότι έχει δίκιο ο εισηγητής γενικότερα. Ο, καθώς και στο ότι θεωρεί ότι είναι υπερβολικά μακρά η διορία που έχει δοθεί και ελπίζω να εγκριθεί το συντομότερο το θέμα. Αν θέλετε μια σύντομη ψηφοφορία αύριο, αν μπορείτε να δεχτείτε ψηφοφορία μαζική. Α, τότε μπορεί να γίνει. Πας κάτω από τους πράσινους. Ναι. Εγώ ήρθα με καθυστέρηση και γι' αυτό θέλω απλώς να χαιρετήσω τη δουλειά, την εξαιρετική δουλειά του συγητή. Εμείς δεν καταθέσαμε τροπολογίες, άρα δεν μπορώ να πω και πολλά. Είμαστε υπέρ της συμβιβαστικής που είναι πολύ καλή και που δεν αδικεί κανέναν. Και το ίδιο θα αντικατοπτριστεί, θα ελπίζω και στη γενικότερη ψηφοφορία το ίδιο πνεύμα. Δεν έχουμε πρόβλημα οι πράσινοι. έχουμε. Έχω εγώ. Είναι πολύ τεχνικό το θέμα αλλά αφορά εκατομμύρια ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα τελεφερίκ και είναι σημαντικό θέμα η ασφάλειά τους. Ξέρω ότι θελήσατε να διασφαλιστεί ότι δεν θα αδικηθεί καμία τοποθεσία με τελεφερίκ που έχει ιστορικές ρίζες κτλ. Ευχαριστώ τον εισηγητή αλλά το ότι κάτι είναι τεχνικό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο σημαντικό από άλλα. Η Ρόζα πάλι. Πολλοί φοβήθηκαν ότι θα καταστούν τα πράγματα δυσκολότερα για τόσους ε, εργάζονται ή έχουν τελεφερήκ. Εμείς θεωρούμε ότι διευκολύνει τα πράγματα η νομοθεσία αυτή και η έκθεση θα ανοίξει την αγορά για εκείνους που παράγουν ανταλλακτικά κλπ. Και δεν θα δυσκολέψει τα πράγματα για όσους λειτουργούν τελεφερικ. Ευχαριστώ λοιπόν και όλους εκείνους που συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάτι να σχολιάσει. Σας ευχαριστώ. Εν γέννη, υποστηρίζουμε τις προτάσεις που έγιναν αποδεκτές από την εισηγητρία, από την εισηγητή και τι συμβαστικέ τροπολογίες. Αν λοιπόν αυτό είναι το μήνυμα του εισηγητή, να ενσωματωθούν οι νέες τεχνικές λύσεις οι οποίες προσφάτως επισημάνθηκαν για όλους μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, έχουμε το πρόβλημα του να συμπεριληφθεί η αρχή της πρόληψης σε τέτοιου είδους νομοθεσία. Γιατί μιλάμε για μια νομοθεσία πλήρους εναρμόνισης ναι. και όλες οι ψυχές ασφάλειας καλύπτονται απόλυτα από τον κανονισμό. Πέρα από την αρχή της πρόληψης. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι οι διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια καλύπτουν όλες τις πτυχές της ασφάλειας και της υγείας και ο κανονισμός δίνει την αρμοδιότητα στις αρχές να αποσύρουν προϊόντα τα οποία δεν είναι ασφαλή από την αγορά, ακόμη και αν φαίνεται ότι συνάδουν με τις διδάξεις του κανονισμού. Άρα όλες οι επιτυχίες της ασφάλειας καλύπτονται απόλυτα από τον κανονισμό και άρα ως εκ τούτου δεν χρειάζεται η αναφορά στην αρχή της πρόληψης. Σας ευχαριστώ πολύ. We don't Δεν ε, θα ξανα... ξανακινήσει γύρος ε, ερωτήσεων από τους κοιόδους και από τους συζητητές. Αν έχετε κάτι μπορείτε να το θέσετε κατευθείαν ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την ιδία. Αν θέλετε να δευτερολογήσετε, πάρτε το λόγο, αλλά εν συντομία παρακαλώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνω τη θέση σας, αλλά με όλον τον σεβασμό θεωρώ ότι δεν συγκρίνεται παρόμοια πράγματα. Λέτε ότι πρόκειται για μέτρα εναρμόνισης και ότι όλα τα, όλες οι πτυχές έχουν προβλεφθεί. Δεν είναι όμως αυτό το ναι. ίδιο οικονομικής άποψης. Με το να αναφέρουμε ότι υπάρχει μια γενική νομική αρχή που τις ξεπερνάει όλες τις διατάξεις. Δεν είναι κατανοώ το επιχείρημα. Θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση κατηδίαν γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση. Μπορεί να υπάρξει πλήρη εναρμόνιση και η αρχή της πρόληψης. Σας ευχαριστώ που το διευκρινίσατε. Ίσως θα μπορούσατε να υποφεληθείτε γιατί είμαστε στην ώρα μας και μάλιστα και πριν από την ώρα μας και η κυρία Στήλη θα πρέπει να φύγει σε λίγο. Ίσως θα μπορούσατε λοιπόν να το συζητήσετε αυτό κατηδίαν με την ε, Επιτροπή. Σα ευχαριστώ. Το επόμενο λοιπόν θέμα στην εμερήσια διάταξη είναι η γνωμοδότηση που καταρτίζουμε για μια ενευρωπαϊκή στρατηγική ενεργειακή ασφάλεια. Η κυρία Φίλη Μενόβα είναι η συγγήτρια. την καθίσταται από την κυρία Κάλλας. Η Καθήλυν αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Βιομηχανία. Θα καταδεχθούν 82 τροπολογίε, τι οποίε και θα συζητήσουμε. Ξέρω ότι δεν έχουν καταστάσει και κάποιοι σκιώδει. Πολύ ωραία. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Κάλλας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Χισμένα μου ζητήσε να σας διαβάσω τα εξή, μια και δεν μπόρεσα, να είναι εδώ πέρα σήμερα. Μετά από προσεκτική εξέταση όλων των τροπολογιών που κατατέθηκαν και σε ό,τι αφορά τι αρμόδιε τη Επιτροπή ΙΜΚΟ, θεωρεί ότι η γνωμοδότηση τελικά αποτελεί το αποτέλεσμα μιας ε, αμοιβαίας συνεργασίας ναι. και αποτυπώνει λοιπόν τι τροπολογίε που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητα τη επιτροπή ΙΜΚΟ για να ολοκληρώσουμε, για να συμπληρώσουμε την γνωμοδότηση και προκειμένου να δώσουμε όλες αυτές τις επιπλέον πτυχές που χρειάζονται. Πέντε συμβιβαστικές τροπολογίες περιλαμβάνονται. Η πρώτη έχει να κάνει με την ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο κατακαιρματισμός της αγοράς, τονίζοντας την ανάγκη πιο ε, σωστής εφαρμογής των ε, διατάξεων του ενεργειακού πακέτου και την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ κρατών μελών. Δεύτερη συμβαστική τροπολογία για το θετικό αντίκτυπο τη ενοποίηση τη αγορά προκειμένου να υπάρχουν πιο σωστέ τιμέ στην ενεργεία. Τρίτη τροπολογία συμβαστική. Τα α, μέτρα ενεργειακή αποδοτικότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι στρατηγικέ επενδύσει ε, συμπεριλαμβανομένου το σύστημα ε, ICT για να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Επόμενη συμβαστική τροπολογία για τις ανανεώσιμες ε, περιφραντικός και οικονομικός αντίκτυπος, το γεγονός ότι αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη μείωση της ενεργειακής ε, ανάγκης. Και τέλος, ε, η διασύνδεση για, ως τρόπος μεγαλύτερης ενεργειακής ασφάλειας. Ε, θεωρεί η συγχύτρια ότι θα είναι χρήσιμη τελική γνωμοδότηση στο έργο τη Επιτροπή Διαμηχανία. Και θα ήθελε εκ νέου να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους και όλους τους υπαλλήλους για τις ε, προσπάθειές τους και για τη συνεργασία τους. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you. Mrs. Κυρία Τούν, εσείς αντικαταστάτε τον Αντώνιο. Μάλιστα. Εγώ θα αντικαταστήσω λοιπόν και πάλι τον Αντώνιο και τιμή μου μεγάλη. Είναι υπεύθυνο από πλευρά μα για την έκθεση αυτή, για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ζητώ συγγνώμη για την απουσία του για μια ακόμη φορά. Ευχαριστεί την εισηγήτρια. Επέδειξε πνεύμα συνεργασίας και όλες οι τροπολογίες του ΕΛΚ έγιναν αποδεκτές. Οι πέντε συμβιβαστικές οι οποίες προτάθηκαν από τον εισήγητη θα υποστηριχθούν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αύριο. Οι συμβιβαστικές αυτές τροπολογίες συνδυάζουν τις ιδέες των μελών της Επιτροπής μας ανεξαρτήτως πολιτικών ομάδων και συνεισφέρουν στην βελτίωση του περιεχομένου ε, της αρχικής ε, ε, διατύπωσης. Ο Αντώνιο του του White πιστεύει ότι και για την ενέργεια θα πρέπει να υπάρξει μια πιο έντονη διατύπωση. Από όλε τις ιδέες που ακούστηκαν, ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα υπογραμμίσει τις εξή. Βασική προϋπόθεση για την δημιουργία της μελλοντικής κοινής αγοράς ενέργειας είναι και το τρίτο πακέτο, και επιπλέον ενεργειακές διασυνδέσεις όπως επίσης και η, η συνέχιση του εξυγχρονισμού του, του δικτύου. Ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χειροκροτά ε, την ε, πρόταση του κυρίου Ιούνκερ για την βελτίωση ναι. της αποδοτικότητας της ενέργειας, ε, προσπάθειες που χρηματοδοτούνται από το νέο στρατηγικό αυτό ταμείο. Τρίτον, είναι πάρα πολύ θετικό για τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και ε, γενικότερα για την οικονομία να διαπιστώσουμε ότι οι πολιτικές μας στον τομέα της ενέργειας αποτελούν στρατηγικού τύπου μακροπρόθεσμες πολιτικές και θα προσελκύσουν επενδύσεις βοηθώντας και τον τομέα των κατασκευών και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Και τελευταία ιδέα, ε, ο κύριος Σίστουρι White θέλει να υπογραμμίσει ε, τον τερματισμό της ύπαρξης των ενεργειακών νήσων. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, διότι θα προσφέρει πολλά στους καταναλωτές που θα έχουν πρόσβαση σε ενέργεια από πολλαπλές πηγές και με καλύτερες τιμές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να σας θυμίσω, λέει η Πρόεδρος, ότι οι καρέκλες που έχουν το όνομα του μέλους μπροστά είναι για τα μέλη μόνο και όχι για τους mm. βοηθούς τους γιατί μας μπερδεύεται και δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποιον θα δώσουμε το λόγο. Λοιπόν, αμέσως βλέπω εδώ ότι έχει έρθει α, ο κύριος Νίλσον. Του δίνω το λόγο. Thank you. It's uh, energy. Uh, Yeah. Ευχαριστώ. Ναι, πώς τι. Τέσσερις μου είχαν πει τέσσερις γι' αυτό, γι' αυτό. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι το θέμα το επεξεργαστήκαμε σε πνεύμα καλής συνεργασίας και σε αναζήτηση συμβιβασμών. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για τη δουλειά του συγκητή. Για την ομάδα μας άλλα θέματα ήταν σημαντικότερα από άλλα βέβαια αλλά αλλά κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Πολλές φορές ξεχνάμε πόσα πολλά μπορούν να γίνουν για αυτό το θέμα. Όταν ήμουν δήμαρχος σε ένα, στο βόρειο τμήμα της Σουηδίας, όπου το κλίμα είναι πολύ ψυχρό, κανονικά θα κόστιζε πάρα πολύ η θέρμανση των σπιτιών. Πριν από 25 χρόνια αρχίσαμε ένα πρόγραμμα με συμβούλους συμβούλους για την αποδοτικότητα. Σε όλη την Σουηδία γινόταν αυτό το πρόγραμμα και με αποτέλεσμα πολλοί ιδιώτες, εταιρείε και τοπικές αρχές να τύχουν αυτών των συμβουλών ως προς το πώς θα μπορούσαν να, να μειώσουν την κατανάλωση και το κόστος και γι' αυτό παρά το ψυχρόν του κλίματος η θέρμανση των οικειών δεν ήταν τελικά πιο ακριβή στο βορρά από ό,τι στο νότο ή στην κεντρική Ευρώπη. Μπορούν λοιπόν να γίνουν πολλά πράγματα εδώ. Αλλά όπως σας είπα είμαι ικανοποιημένο από τη δουλειά του εισηγητή και είναι πολύ καλή η έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Βίκυ και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έκανε σε ό,τι αφορά τι συμβαστικέ τροπολογίε. Όντως καταφέραμε, όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι, να βρούμε μια ευρεία συνένεση για τα όρια του καθενός πέρα από τα όρια των ομάδων. Αυτό είναι σημαντικό ασφαλώς για όλους, για όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς θα ψηφίσουμε και τις τροπολογίες που δεν μπήκαν στους συμβιβασμούς, αλλά συμφωνούμε επί της κοινής βάσης και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνω ότι υπάρχει ομοφωνία σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα. Όσο πιο λίγη ενέργεια χρειαζόμαστε και καταναλώνουμε, τόσο λιγότερο εξαρτημένοι θα είμαστε και από άλλες ναι, ναι. χώρες και τόσο καλύτερο θα είναι αυτό και για τους πολίτες σε ό,τι αφορά το κόστος της ενέργειας. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο. Είναι καλό το ότι υπάρχει έκκληση για νομική βεβαιότητα και εγγύηση σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σίγουρα θα μας απασχολήσει αυτό και στη μελλοντική ναι, έκθεση και γνωμοδότηση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σταθερό κλίμα, μια σταθερή ατμόσφαιρα σε ό,τι αφορά την νομική, τις νομικές διατάξεις και Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά θα έκανε να μην αλλάζει τέτοιε διδάξει κάθε και λίγο. Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι τον εισηγητή, του κοιόδη και του βοηθού του πάντα. Δεν είναι εδώ ο κύριος Μαστάλκα. Η κυρία Ντουραν. Ο κύριος Ντουραν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το είπαν οι προλαλήσαντες. Μιλάμε για την ενέργεια, μιλάμε για την διασφάλιση της ε, προμήθειας ενέργειας. Είναι μια ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να φανεί εδώ ικανή και χρήσιμη. Η αποδοτικότητα της ενέργειας είναι πολύ σημαντικό θέμα, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά ε, και για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων γιατί μπορεί να βοηθήσει ε, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ενέργειας για συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε το θέμα της αποδοτικότητας και για την καταπολέμηση των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον τομέα της οικολογίας. Δεν θα επανέλθω στα θέματα τώρα της ασφάλειας και της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν και αυτά μεγάλη σημασία. Αυτά ήταν μια εισαγωγή. Να πω ότι η δουλειά που έγινε είναι μια εξαιρετική δουλειά. Δείχνει ότι η εισηγήτρια ότι θέλει να υπάρξει μια συνένεση και γι' αυτό θα υποστηρίξουμε τις πέντε συμβιβαστικές προτάσεις. Είναι σαφές ότι υπάρχει επιθυμία να βρεθεί μια κοινή λύση Υπάρχει ένα σημείο όμως πάνω στο οποίο δεν ξέρω αν ο εισηγητής το έχει παραβλέψει ή αν υπάρχει μια διαφορετική σκοπιμότητα η οποία μου διαφεύγει. Εμείς μέσω της τροπολογίας 47 ζητήσαμε να υπενθυμηθεί ότι η αποδοτικότητα αυτή έχει θετικά αποτελέσματα στην κατάρτιση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και θετικά αποτελέσματα για τις μικρομεσαίες. Αυτό δεν έγινε δεκτό. Γιατί αυτό δεν συμφωνείτε με αυτό. Πιστεύω ότι συμφωνείτε. Θα ήθελα εφόσον αυτό είναι εφικτό να προσθεθεί εκ νέου το τμήμα αυτό της τροπολογίας μας σε 47, έστω και μέσω ψηφοφορίας, ως προσθήκη στη συμβιβαστική. Αυτή είναι η μοναδική παρατήρηση. Κατά τα άλλα υποστηρίζουμε τις πέντε προτάσεις. Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα ήθελε το λόγο. Όχι λέει η κυρία Φόρντ. Λοιπόν σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Και πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερα σε θέματα καταναλωτών όσο περισσότερες αρμοδιότητες συγκεντρώνουμε στο εσωτερικό της Επιτροπής μας τόσο το καλύτερο. It's because we are the committee that looks at things from the consumer as well as from the internal market perspective. And the consumer perspective on these issues is really important as well. So thank you very much for... Η σημασία λοιπόν και αυτό για τις αρμοδιότητες Επιτροπής μας. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στη συνέχεια στο 8 την ε, γνωμοδότηση για την προστασία των λεγόμενων εμπορικών μυστικών. Η Λάουρα Κόμη είναι η συγγήτρια. 211 τροπολογίες έχουν κατατεθεί στην έκθεση αυτή. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η συγκεκριμένη έκθεση. Δίνω το λόγο λοιπόν στην κυρία Κόμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν είναι παρηγορητικό στο ότι στη νομική επιτροπή οι τοπολογίες είναι περισσότερες. Σήμερα λοιπόν θα αξιολογήσουμε τις συμβιβαστικέ τροπολογίες για να δούμε αν μπορούμε πράγματι να εξισορροπήσουμε τα, ε, ε, τα συμφέροντα που ε, εδώ διασταυρώνονται. Υπάρχουν 23 συμβιβαστικές τροπολογίες. Θα προσπαθήσω να τις διατρέξω με συνοπτικό τρόπο. Η πρώτη συμβιβαστική τροποποιεί την αιτιολογική 8. Από τη μία μιλάει για την ελάχιστη εναρμόνιση και από την άλλη για την δυνητική παρούσα ή δυνητική εμπορική αξία και τεχνογνωσία. Συνάδελφος Ντουράν και αυτό άπτεται και τη συμβιβαστικής 9 σχετικά με το άρθρο 2. Η δεύτερη ε, συμβιβαστική εισάγει ένα νέο 10. Αναφέρεται η ανάγκη σεβασμού των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του ρόλου των συλλογικών συμβάσεων. Είναι κάτι το οποίο έθεσαν οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι. Δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να περιληφθεί στο ρυθμιστικό κομμάτι, είναι κάτι που ισχύει για ορισμένες χώρες οι οποίες ε, ε, θέτουν σε λειτουργία και εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά όχι σε όλες τις χώρες. Μπορούμε να το βάλουμε όμως στην αιτιολογική σκέψη. Η τρίτη συμβιβαστική εισάγει την βασική αρχή σύμφωνα με την οποία τα εμπορικά μυστικά δεν θα πρέπει ο σεβασμός τους να οδηγεί στην παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών, των εργαζομένων και στις συνδικαλιστικές τους ελευθερίες. Αυτά τα σημεία που έχουν θέσει οι γκουε, οι πράσινοι και οι σοσιαλιστές γίνονται ε, δεκτές. Και δεν υπάρχει απλά γενική αναφερά στο ε, το γενικό συμφέρον. Ζητήθηκε από την κυρία Κόμη να ομιλεί πιο αργά. Λοιπόν, η πέμπτη συμβιβαστική ε, διαγραφή ε, στα τρία χρόνια για την προστασία των ε, συγκεκριμένων αυτών εμπορικών απορρίτων. Η Επιτροπή είχε ζητήσει ένα με δύο χρόνια, κάποιοι είχαν ζητήσει έξι χρόνια, νομίζω ότι τα τρία χρόνια είναι μια καλή συμβιβαστική λύση. Και αυτό ε, περιλαμβάνεται και στη συμβιβαστική 15. Η πέμπτη συμβιβαστική ότι λέει, λέει ότι το εύρος ε, εφαρμογής αναφέρεται σε εμπορικά απόρριτα και προϊόντων και υπηρεσιών και εδώ έχει κατατεθεί μια τροπολογία που ορίζει καλύτερα τις υπηρεσίες έτσι ώστε να διαπιστώνονται οι παραβιάσεις όπου αυτές υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό το ειδικό χαρακτηριστικό νομίζω ότι θα πρέπει να ενταχθεί μόνο στην αιτιολογική σκέψη και όχι στο διακανονιστικό νομικό δεσμευτικό κομμάτι. Λοιπόν, η έκτη περιλαμβάνει ένα καλύτερο ορισμό και μια καλύτερη περιγραφή του λεγόμενου εμπορικού απορρίτου. Η έβδομη συμβιβαστική συγκεκριμενοποιεί ένα σημείο το οποίο κρίνουμε πάρα πολύ σημαντικό. Το πανάρωμα που έχουμε μπροστά μας είναι, ε, χαρακτηρίζεται από πολυδιάσπαση και υπάρχουν σε ορισμένες χώρες ε, κανόνες πολύ πιο αυστηροί. Από τη μία λοιπόν υπάρχει ανάγκη ε, να καθοριστούν κοινοί κανόνες, αλλά από την άλλη εκεί όπου υπάρχουν σωστοί κανόνες και ισχυρότεροι δεν θα πρέπει να αμφισβητηθούν. Πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει μια βελτίωση συνολικά της νομοθεσίας. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Η ενδέκατη αναφέρεται στο ότι η χρήση του εμπορικού απορρίτου ε, μπορεί να είναι παράνομη όταν αυτός που το χρησιμοποιεί ε, το κάνει με παράνομο απλά τρόπο. Η δωδέκατη απόκτηση, η χρήση και η κυκλοφορία του εμπορικού απορρίτου είναι νόμιμη εφόσον καλύπτεται από το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο και χρησιμοποιείται κυρίως από τον ε, δημόσιο τομέα. Η 13η συμβιβαστική ξεκαθαρίζει το κείμενο σε επίπεδο διατύπωσης και δεν θα καθυστερήσω γι' αυτό. Η 16η αναφέρεται στο ότι η υποχρέωση εμπιστευτικότητας αποφασίζεται ή μπορεί να μην εφαρμοστεί εφόσον υπάρξει μια δικαστική απόφαση σε τελικό στάδιο. Αυτά πάντα για το άρθρο 2. Όπως είπα στην αρχή η 16 η συμβιβαστική αναφέρεται στο άρθρο 2. Η 17η. Εδώ πάντα τίθεται το θέμα της εμπιστευτικότητας και οι υπόλοιπε συμβιβαστικέ προτάσεις βελτιώνουν τη διατύπωση του κειμένου και δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα. Να προσθέσω ένα θέμα το οποίο έχω αφήσει σε εκκρεμότητα. Το θέμα της κατανομής των αρμοδιοτήτων για την απόκτηση, χρήση και παράνομη μάλιστα χρήση του εμπορικού απορρίτου. Νομίζω ότι η ευθύνη θα πρέπει να είναι αντικειμενικά καθορισμένη. Αυτή είναι η καλύτερη λύση να πω στους συναδέλφους της φιλελεύθερης ομάδες ότι decidiamo di valutare Ότι το θέμα της αμέλειας ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ειδικά εδώ να ξεχωριστεί από τα υπόλοιπα θέματα. Ξαναζητήθηκε από την κυρία Κόμη να ε, μην ομιλεί γρήγορα. Λοιπόν, ή εμείς θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε υποκειμενικά το θέμα της ενοχής ή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε βάρος μόνο στις ρυθμιστικές αυτές προτάσεις. Εγώ είμαι υπέρ ε, της, ε, ε, του αντικειμενικού τρόπου μετακήρυσης. Το θέμα δεν είναι το ποια είναι η αιτία η οποία οδήγησε στη βλάβη. Το θέμα είναι η σωστή αξιολόγηση της ίδιας της βλάβης. και νομίζω ότι μίλησα βέβαια αρκετά, νομίζω ότι μίλησα γρήγορα, ίσως γιατί ένας από τους κοιόδης είναι και αυτός Ιταλός. Πράγματι μας βοηθήσατε, αλλά προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε κάποιες τεχνικές ρυθμίσεις και κάποιους αριθμούς. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πάρα πολύ χρόνο και κάνατε μια τεράστια προσπάθεια. Ευχαριστώ κύριε Ακόμη. Ο κύριος Κοφεράτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Γενικά οι Ιταλοί όταν ομιλούν, ομιλούν οργά. Εγώ είμαι εξαίρεση, από μένα μη φοβηθείτε. Μετά από τη συνάντηση των σκιωδών, πριν λίγες εβδομάδες, πήραμε τις συμβιβαστικές προτάσεις, πήραμε τις 23 λοιπόν αυτές τροπολογίες, τις οποίες παρουσίασε η συνάδελφος Κόμη Σήμερα το πρωί η σοσιαλιστική ομάδα, στη σοσιαλιστική ομάδα και η συγγήτρια και οι υπόλοιποι σκιώδεις απέστειλαν κάποιες παρατηρήσεις σε όλες τις συμβιβαστικές προτάσεις οι οποίες έγιναν. Εμείς εκτιμούμε δεόντως την προσπάθεια την οποία έκανε η συνάδελφος. Θα πρέπει όμως να τονίσω ότι η ομάδα μου θεωρεί ότι τα πιο σημαντικά θέματα για μας, για τους σοσιαλιστές, ή δεν καλύπτονται, δεν έχουν επιληθεί δηλαδή τα προβλήματα τα οποία έχουμε, ή έχουν ε, επιληθεί μόνο ε, επιμέρους, δηλαδή έχουμε ένα ευρύτατο πεδίο διαφωνίας. Είχαμε επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι για μας τα πιο σημαντικά πεδία είναι τέσσερα και θα ήθελα με συντομία να σας τα παρουσιάσω. Το πρώτο αφορά την ανάγκη έκφρασης με μεγαλύτερη ευκρίνεια και καθαρότητα ότι το know-how και οι επαγγελματικές εμπειρίες των εργαζομένων δεν μπορούν να θεωρηθούν εμπορικό απόρριτο. Και αυτό από τις συμβιβαστικές προτάσεις δεν διαφαίνεται. Δεύτερον, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε με καλύτερο τρόπο την επικράτηση πάντα και την προτεραιότητα του γενικού συμφέροντος και των δράσεων της δημόσιας διοίκησης γενικότερα. Τρίτον, θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα επακριβέστερο ορισμό της έννοιας του εμπορικού μυστικού, του εμπορικού απορρίτου και της παράνομης χρήσης του. Η συμβιβαστική πρόταση η οποία έγινε δεν μας καλύπτει εδώ. Ένα τέταρτο ε, γενικό σημείο διαφωνίας αναφέρεται στην ε, μη τήρηση του σεβασμού της ελευθερίας έκφρασης και του καθήκοντος ενημέρωσης και έκφρασης. Να κάνω τώρα κάποιες πολύ σύντομες ε, πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Θα πω σαν παράδειγμα στο σημείο 2 δεν λαμβάνεται υπόψη το αίτημά μας της εισαγωγής της έννοιας της εμπορικής αξίας και του οικονομικού συμφέροντος. Όπως επίσης και στο άρθρο 3, στα πλαίσια της συμβιβαστικής πρότασης δεν λαμβάνονται υπόψη κάποιες τροπολογίες σημαντικές όπως η 93, η 109, η 110, που αναφέρονται στην παράνομη απόκτηση για οικονομικά κέρδη ε, mm. τέτοιου είδους απορρίτων. Και εδώ τίθεται το θέμα της εμπλοκής του εργαζομένου με αντικειμενικό τρόπο και χωρίς ε, βλέψεις παρανομίας. Η διατύπωση του άρθρου 4 θα πρέπει να αλλάξει λοιπόν γιατί δεν περιλαμβάνονται τροπολογίες όπως οι 121 και 122 που αφορούν την εξαίρεση πληροφοριών από τους, ε, από τους εργαζομένους, όπως επίσης και της εξαίρεσης της έννοιας του γενικού συμφέροντος, καθολικού συμφέροντος. Επίσης έχουμε ένα θέμα με τις τροπολογίες 4 και 5. Υπάρχουν μικροδιαφωνίες και σε άλλα σημεία Έχουμε εδώ κάποια προβλήματα με τη μορφή του κειμένου. Αλλά εγώ παραμένω αν θέλετε στις κομβικές διαφορές τις οποίες υπογραμμίζουν οι τροπολογίες που καταφέσαμε. Και θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια να μας πει εάν θα ήταν χρήσιμο στην παρούσα φάση να αναβληθεί η ψηφοφορία η οποία στην αρχή είχε προβλεφθεί για την επόμενη εβδομάδα. Αν γίνει κάτι τέτοιο ε, θα έλεγα ότι θα έχουμε κάπως περισσότερο χρόνο για να προσπαθήσουμε να γυπνιάσουμε τις ε, ε, διαφορετικές μας απόψεις. Έτσι θα υπάρξει χρόνος για συζήτηση και φοβάμαι ότι μόνο μέσω του χρόνου αυτού θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιες επιπλέον συμβιβαστικές λύσεις. Αν επιβεβαιωθούν οι προτάσεις αυτές αν δεν γίνουν δεκτές οι προτάσεις αυτές φοβάμαι ότι θα περάσουμε αύριο σε ψηφοφορία με τεράστιες διαφορές μεταξύ μας. Να ακούσουμε όλους τους κύριους για να ακούσουμε τα σχόλια. Σε ό,τι αφορά το αίτημα για την αλλαγή της ψηφοφορίας, ανησυχώ, ανησυχώ κάπως. Ανησυχώ. Γιατί όσα γίνονται στη γραμματεία κατά τη διάρκεια του Πάσχα ενδεχομένως να τους δυσκολέψουμε αν αλλάξει η ψηφοφορίας. Για την ομάδα του ECR, η κυρία Μακλάκνη, το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την συγγήτρια για τη δουλειά που συνεχίζει να κάνει για αυτή την ε, γνωμοδότηση. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι να αποτυπώνεται η ανάγκη των επιχειρήσεων να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να προστατεύουν την τεχνογνωσία τους σε οποιοδήποτε κλάδο και να δραστηριοποιούνται. Αυτό τι σημαίνει ότι ο ορισμός του εμπορικού απόρριτου είναι εξαιρετικά σημαντικός και χαίρομαι που προσπαθούμε να αποτυπώσουμε στις τροπολογίες 6 έως 10 τη σημασία αυτή. Κάτι άλλο που με απασχολεί ιδιαίτερα, η προστασία των εμπορικών απορρίτων κατά τη διάρκεια των δικαστικών αγωγών και χαίρομαι που στην τροπολογία 17 αποτυπώνεται αυτό. Η τροπολογία αυτή ταιριάζει και με την δική μου τροπολογία, αλλά το πρόβλημά μου εξακολουθεί να είναι η περίοδος απρεβισμού και θα προσπαθήσω να την ε, μεγιστοποιήσω. Πιστεύουμε ότι πραγματικά θα ωφελήσει το γεγονό ότι θα υπάρξει μια πιο μεγάλη τέτοια περίοδο, ιδιαίτερα για περιπτώσει που είναι πάρα πολύ τεχνικέ, όπου ε, η προετοιμασία διαρκεί χρόνια ολόκληρα. Και πραγματικά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει επαρκή περίοδο. Αν ε, περιοριστεί αυτή η περίοδο περιορισμού, ουσιαστικά θα ρίχνουμε τον κόσμο να πάρουν ε, κοντόφθαλμα μέτρα, όπως για παράδειγμα δικαστικές αγωγές. Μπορεί να μην ε, να μην ε, χρησιμοποιήσουν τον χρόνο που χρειάζεται για να διαπιστώσουν ότι στην πραγματικότητα δεν χρειαζόταν αυτή η αγωγή. Να κοιτάξουμε λοιπόν την τροπολογία 15 που θεωρώ ότι δεν είναι αποδεκτή από την ομάδα μας, αλλά είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την εισηγήτρια για να καταλήξουμε σε έναν λογικό συμβιβασμό. Να διασφαλίσουμε επίσης ότι όταν νομοθετούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μειώνουμε τα προϊόντα, δεν χρησιμοποιούμε προστασία για κάποια εμπορικά απόρριτα το, η μείωση της περίοδου περιορισμού σημαίνει λιγότερη προστασία και το δεν τίθεται σε μεν, αλλά να ληφθούν υπόψη οι προσωπικές μας προτεραιότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και προσβλέπουμε στη συνεχιζόμενη συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Κάλλας από τους φιλεύθερους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για, τις, ε, για τους συμβιβασμούς. Αλλά μου φαίνεται ότι έγινε κάποια συνεδρίαση μεταξύ των σκιωδών της Ιταλικής Αντιπροσωπείας γιατί ο σκιώτης των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών αναφέρθηκε σε μια συνεδρίαση όπου συζητήθηκαν οι συμβαστικές τροπολογίες. Εγώ δεν ε, προσκαλέστηκα σε οποιαδήποτε τέτοια συνεδρίαση. Την προηγούμενη εβδομάδα τις είδαμε τις τροπολογίες αυτές τι συμβαστικές, αλλά δεν είδα να είχαμε ευκαιρία να τις συζητήσουμε μεταξύ των ε, σκιωδών, όπως και να έχει. Κάποιες συμβαστικές ενδεχομένως να τις υποστηρίξουμε. Για κάποιες άλλες έχουμε ανησυχίες. Στη συμβαστική τρία συμφωνούμε με την ε, στάση της εισηγήτριας να καταγραφούν τα δημόσια συμφέροντα τα οποία θα πρέπει να εξασφαλιστούν και να υπάρχει σαφήνεια στον κατάλογο εξαιρέσεων στο, στο, στον άρθρο 4. Στο άρθρο 4 αυτό όμως θα δοθεί στην Επιτροπή ως έχει. Τι θα γίνει. Χαίρομαι επίσης που η συγγήτρια διευκρινίζει τις υπηρεσίες της τελογικής σκέψης. Στα 17, στην τελογική σκέψη 17 η τροπολογία 52 που κατέφτασε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Όσο αφορά τώρα την περίοδο απεριορισμού, μας ε, απασχολούν οι μεβαστικές λύσεις. Υποστηρίξουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των δύο χρόνων ένα σχόλιο τώρα για αυτό που είπε η εκπρόσωπος ε, του ECR για τις κυρώσεις. Το επιχείρημά σας είναι κατά τον, ε, της μεγαλύτερης περίοδου περιορισμού, γιατί αυτό θα περιορίσει τις δραστηριότητε των ε, επιχειρήσεων για την ελάχιστη εναρμόνιση. Το είπα και πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν υποστηρίζω τη συμβαστική 7 για την δυνατότητα των κρατών μελών να εισαγαγούν πιο πολλά προστατευτικά μέτρα. Θα, προστα... θα προτιμούσα να το 2, 3 και 7 να εναρμονιστούν σε ό,τι αφορά τον ορισμό του τι είναι νόμιμο, τι είναι παράνομο και την περίοδο περιορισμού και αυτή πρέπει να εναρμονιστεί. Γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, αν ο στόχος μας είναι να έχουμε ενιαίους ε, κανόνες, επειδή άλλως είναι πολύ δύσκολο οι επιχειρήσεις να καταλάβουν πού ισχύουν και πώς ναι. ισχύουν οι διαφορετικοί κανόνες, αυτά τα σημεία θεωρώ ότι θα πρέπει να εναρμονιστούν. Τα διαδικαστικά, ναι, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν εδώ διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες και να παραμείνουν. Εκεί λοιπόν μπορεί να υπάρχει κάποια ε, ευελιξία για την συμβαστική 10 για τον ορισμό της παραβίασης των προϊόντων που παραβιάζουν. Συμφωνώ ότι υπάρχει σύγχυση, τι σε ό,τι αφορά την αντίστροφη μηχανική, το reverse engineering, την αναφορά στα δημόσια, δημόσιες υπηρεσίες. Αν θέλουμε να γίνει αυτή η αναφορά, προτιμώ τον ορισμό που έχει γίνει στην τροπολογία 36. Η αναφορά στο εθνικό δίκαιο, λίγο από το πριν το άρθρο 4, που αναφέρει τις εξαιρέσεις και την αποκάλυψη απορρίτων, θεωρώ ότι μάλλον προκαλεί τη μεγαλύτερη σύγχυση στην ε, τροπολογία 18. Είναι σημαντικό να αποδειχθεί ότι υπήρχε ε, απόρριτο επιχειρηματικό το οποίο όντως αποτελούσε τέτοιο και μετά το δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον όντως υπήρχε αυτό το εμπορικό απόρριτο. Δεν μπορούμε αυτό να το ρυθμίσουμε με την οδηγία. Και να μην μπαίνουμε στα νερά των δικαστηρίων, να τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μπορεί να υπάρχει λοιπόν επαρκής βαθμός ασφάλειας και βεβαιότητας. Κοιτάξτε την ε, τροπολογία 190 της Άλντε με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Θα αποστείλουμε τις, ε, τα σχολιά μας και ίσως μετά θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε σε συνάντηση των σκιωδών. Ο κύριος Κομφεράντη και η κυρία Δεν νομίζω ότι θέλουν να διευκρινίσουν ότι δεν έχει γίνει τέτοια συνάντηση. Να σας καθησυχάσω. Η συνάντηση αυτή έγινε πριν δύο εβδομάδες. Εσείς ήσασταν εκεί, εγώ δεν ήμουν. Είχα ένα ιδιωτικό πρόβλημα που με εμπόδισε να πάρω μέρος. Δεν έχει υπάρξει καμία Ιταλο-Ιταλική συνάντηση σεβαστήκαμε πάντα τους κανόνες και οι πολιτικές αποστάσεις ε, ανάμεσα στις θέσεις της κόμη και τις δικές μου είναι τεράστιες και απαγορεύουν άμεσες επαφές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαστάλκα δεν είναι εδώ. Ο Πασκάλ τώρα είναι από Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρίτη φορά παίρνω το λόγο. Πρωτοφανές. Είχα ήδη πει την προηγούμενη φορά ότι είχα το δυσάρεστο συνέστημα για την έκθεση αυτή ένα δυσάρεστο συνέστημα όχι για τη δουλειά της συζητηρίας αλλά για το πνεύμα της η νομοθεσία για τα εμπορικά μυστικά ή για το εμπορικό απόρριτο στόχευε στην προστασία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν τη δυνατότητα όπως οι μεγάλες να προστατεύσουν τα μυστικά τους. Αυτό δεν μου δημιουργεί πρόβλημα. Αρχικά το είχα πει και στην Επιτροπή. Υπά, θεωρούσα ότι υπάρχουν ήδη προστασίες από τα κράτη-μέλη. Αλλά τέλος πάντων ας δεχτούμε ότι στα πλαίσια της μιας γενικευμένης προστασίας, επειδή μερικές χώρες δεν έχουν, προβλέπουμε αυτά. Αυτό το δέχομαι. Αυτό που με ενοχλεί και με ανησυχεί είναι ότι φοβάμαι ότι το κείμενο αυτό για το εμπορικό απόρριτο δεν χρησιμοποιείται πια για τον αρχικό του στόχο αλλά ευνοεί τις μεγάλες φαρμακευτικές ιδίως εταιρείε που παραχωρούν την, μετά από μερικά χρόνια κανονικά την άδειά τους για να δημιουργηθούν γενώσιμα αλλά ότι με αυτή την νομοθεσία θα έχουν την ικανότητα λόγω του δίθεν εμπορικού μυστικού ή απορρίτου να μην το πράττουν στο εξή. Αυτό με ανησυχεί. Και ο μόνος τρόπος να, να με καθησυχάσετε θα ήταν εάν υπάρχει βέβαια τέτοια κακή πρόθεση θα ήταν να παραμείνουμε στην αρχική λογική που είχε προσπαθήσει να την εξωσορροπήσει η Κομισιόν. Βλέπω όμως ότι το αντίθετο τελικά γίνεται. Δηλαδή Αντί να περιορίζουμε μέσω ενός αυστηρότερου ορισμού τι είναι το εμπορικό απόρριτο αποκλείοντας συγκεκριμένα ότι δεν πρέπει να καλύπτεται από αυτό, ότι αντιτίθεται στα δικαιώματα και στην κινητικότητα των εργαζομένων πούμε ή στη δυνατότητα να χορηγούν πληροφορίες ορισμένοι πληροφοριοδότες, όλα αυτά πρέπει να εξαιρούνται. Καταρχήν γιατί υπάρχουν άλλα κείμενα οδηγίες, η εθνική νομοθεσία επικουρικά που τα καλύπτουν. Αντί για αυτό όμως η έκθεση είναι τόσο ασαφής που έχουμε το αίσθημα ότι οτιδήποτε μπορεί να συμπεριληφθεί υπό την έννοια εμπορικό απόρριτο όπως κοινωνικά θέματα κλπ. κλπ. Ας μην υπησέλθω σε λεπτομέρειες των τροπολογιών αλλά εάν δεν συμφωνούμε για τον λόγο για τον οποίο πρέπει να υπάρχει αυτό το νομοθέτημα, τότε δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κανένα συμβιβασμό, πράγμα που θα ήταν λυπηρό. Διότι είναι πάντα δυνατόν να πετύχουμε συμβιβασμούς. Δεν θα σας διαβάσω τώρα για να μην σας κουράσω τις τροπολογίες, τις ξέρει και η συγγήτρια, μπορούμε να τις ξαναδούμε, αλλά γενικά υπάρχει εδώ ένα η ανάγκη να επανέλθουμε στην αρχική έννοια του εμπορικού απορρίτου την προστασία δηλαδή συγκεκριμένων διαδικασιών παραγωγής και να αποκλειστεί οτιδήποτε εμποδίζει την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών και καταναλωτριών. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μήπως η Κομισιόν θέλει να προσθέσει τίποτα. Ο κύριος Γκονζάλης. Αι, αι, αι, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έρχομαι Γκονζάλης αλλά σ' άλλες. Η Κομισιόν θέλει απλώς να ευχαριστήσει την Επιτροπή σας για τις συζητήσεις της που τις παρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον, ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και ελπίζουμε το αποτέλεσμα να συμβάλλει και αυτό στην ε, βελτίωση της αρχικής πρότασης. Μερικά σχόλια, αν μου το επιτρέπετε. Πρώτον, η πρόταση δεν δημιουργεί κανένα αποκλειστικό δικαίωμα σε πληροφόρηση, δεν περιορίζει δηλαδή την πληροφόρηση. πληροφόρηση που χορηγείται αυτή τη στιγμή σε οποιονδήποτε μπορεί να συνεχίσει να χορηγείται. Δεν περιορίζει η οδηγία ούτε την ανεξάρτητη λεγόμενη ανακάλυψη ή αποκάλυψη. Κατατέθηκαν πολλές τροπολογίες, δεν συμπεριλήφθηκαν όλες τις συμβιβαστικές, αλλά μερικές περιορίζουν τις ελευθερίες που ανέφερα και πρέπει ίσως να το ξανασκεφτούν οι συντάκτες των Η προτινόμενη οδηγία δεν αλλάζει τους κανόνες που υποχρεώνουν στη χορήγηση πληροφόρησης του κοινού από εταιρείε. Δεν είχαμε σκοπό να περιορίσουμε τους κανόνες αυτούς το εύρος τους. Και τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η πρόταση, την πρόταση θεωρούμε ισορροπημένη και χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό. Όταν η Κομισιόν είχε κάνει την αρχική της παρουσίαση της πρότασης, είπατε με μεγάλο σθένος ότι ένας λόγος για τον οποίο δεν εμπορεύονται μεταξύ τους οι επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά είναι γιατί φοβούνται την αποκάλυψη των εμπορικών τους μυστικών και ότι σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν καμία προσφυγή. Αυτή η πρόταση στόχευε λοιπόν στον, στην προστασία τους. Αν υπήρχε καμία παρατυπία. Προστασία λοιπόν του εμπορικού απορρίτου και όχι τι είναι και τι δεν πρέπει να είναι μυστικό. Θυμάμαι ότι η Κομισιόν τα είχε πει πολύ στεναρά. Οι επιχειρήσεις δεν εμπορεύονται καμιά φορά επειδή φοβούνται με τρίτες χώρες, μεταξύ χωρών, τι θα γίνει για την περίπτωση που παραβιάζονται τα εμπορικά των απόρριτα. υπενθυμίζω δε στους συναδέλφους ότι επειδή μια τροπολογία δεν συμπεριλαμβάνεται σε ένα συμβιβασμό δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα ψηφιστεί κιόλα. Θα ψηφιστεί. Πολλές τροπολογίες καλύπτονται από τις συμβιβαστικές αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τις ψηφίσουμε και εκείνες αλλά μόνο τις συμβιβαστικές. Όχι θα ψηφίσουμε και τροπολογίες που δεν είναι στο συμβιβασμό. Ευχαριστούμε λοιπόν. Δώσαμε τη δυνατότητα στον εισηγητή να αλλάξει την ημερομηνία για την ψηφοφορία στην 23η Απριλίου. Την εισηγήτρια. Αλλά βέβαια ελπίζουμε να γίνεται αυτό, θα τα κανονίσει αυτά η γραμματεία μπορεί να μην γίνεται λόγω πίεσης χρόνου. Θα μας τα πει, θα τα δει η γραμματεία λόγω της πράσινης εβδομάδας του Πάσχα. Οι επιτροπές που ασχολούνται, που είναι αρμόδιες για την εσωτερική αγορά, μπορεί να θέλουν και αυτές να υψώσουν τη φωνή τους και θα οργανωθούν κοινές ψηφοφορίες, η νομική κυρίως επιτροπή. Πάλι η Λάουρα Κόμε τώρα. Εκτός αν η Κομισιόν έχει τίποτα να προσθέσει. Όχι, όχι, όχι. Η Λάουρα λοιπόν. Τώρα για την ημερομηνία, όπως ε, εμείς σαν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουμε τις ημερίδες μελέτης, δεν ξέρω αν μπορούμε να συμπέσουμε για την μικρή αναβολή για την ψηφοφορία θα συμφωνήσω. Για να μπορέσουμε να βρούμε τις καλύτερες ε, διατυπώσεις ε, ε, και δεν είναι στόχος μου η μεγάλη πλειοψηφία το να νικήσουμε αλλά θέλουμε ένα πραγματικά εμπεριστατωμένο κείμενο. Να διαβεβαιώσω ότι συνάδελφο ο κύριος Κοφεράτη ε, δεν συμφωνεί με το κόμμα του που τον έχει εγκαταλείψει. Οπότε πόσο μάλλον με το δικό μας κόμμα. Δεν υπήρξε καμία συνάντηση ιδιωτική μεταξύ μας. Ο διάλογος είναι ανοιχτός και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ε, κοινωνικό. Το θέμα δεν είναι τυπικό. Ε, τώρα κάποιες γενικές παρατηρήσεις μετά από αυτά τα οποία υπόθηκαν για την κινητικότητα των εργαζομένων δεν περιλαμβάνεται μόνο στην αιτιολογική σκέψη αλλά και στα άρθρα. Αυτό το πήραμε από τους σοσιαλιστές και το εκτιμήσαμε. Το άλλο το θέμα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία έκφρασης. Εμείς έχουμε υιοθετήσει πάρα πολλά από τα σημεία τα οποία αρχικά είχαμε δυσκολευτεί να αποδεχθούμε. Είχαμε κάνει κάποιες πρώτες προτάσεις τώρα για τις προτάσεις και του Ντουιράν και του Κοφεράτη που ήταν οι πλέον θα έλεγα διαφορετικές εμείς πετύχαμε ε, να τις εντάξουμε όλες ε, στην αιτιολογική σκέψη. Αν θέλετε να τα εντάξουμε και στο κομμάτι το διακανονιστικό τότε θα το μελετήσουμε εκ νέου. Το θέμα το οποίο εδώ μας απασχολεί είναι η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Μιλάμε για ανάπτυξη Κάνουμε προτάσεις για επενδύσεις, προγράμματα Juncker και μιλάμε ε, για ένα πλαίσιο προστασίας μεν αλλά και αύξησης της γραφειοκρατίας δε. Βασικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε τον πολίτη, να προστατεύσουμε τον δημιουργικό εργαζόμενο που έχει τις συγκεκριμένες ιδέες και από την άλλη να υπάρξει μια κατελάχιστον εναρμόνιση. Αν μια χώρα είναι ικανή ε, να σεβαστεί υψηλότερους κανόνες, αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας εμπνεύσει, αλλά όχι να μας οδηγήσει σε βήματα προς τα πίσω. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τη γραμματεία που έχει επιδείξει ιδιαίτερη ε, ε, υπομονή έτσι ώστε να βρει μια ημερομηνία για την ψηφοφορία που να ταιριάζει και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Θα κοιτάξουμε μια άλλη ημερομηνία, αλλά αν τυχόν δεν βρούμε θα εμείνουμε στην επόμενη εβδομάδα. Πάμε κάπως πιο γρήγορα από ό,τι προεβλέπαμε. Ε, ζητώ συγγνώμη για την αναταραχή. Περνάμε τώρα στο σημείο 10. Για όσους δεν με ακούσατε, θα μιλήσουμε για το 10 πριν το 9. Ελπίζω να μπορέσουμε να τα κλείσουμε τα θέματα αυτά στις 5.30. Έτσι ώστε η συγγήτρια να μπορέσει να πάει στην αντιπροσωπεία, να πάρει το αεροπλάνο μάλλον για να πάει την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, το 10. Γνωμοδότηση για την εφαρμογή της οδηγίας εναρμόνισης τμήματων πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι για γνωμοδότηση στην έκθεση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων βασικός εισηγητής ε, είναι ο κύριος Ρέντα. Είναι όμως εδώ ανάμεσά μας. Έχουν κατατεθεί 82 τροπολογίες και θα δώσω το λόγο στην Κάθριν Στάιλερ για να σχολιάσει αυτές τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και ελπίζω να είμαι σύντομη. Να ευχαριστήσω τους Κιώδης για την πολύ παραγωγική συνάντησή μας την προηγούμενη εβδομάδα για τις 82 αυτές τροπολογίες περιορισμένος αριθμός ε, σε σχέση με τις 550 τροπολογίες της Jillian. Ε, ελπίζω λοιπόν οι συνάδελφοι είναι λίγο πιο ήπιοι μαζί μου. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Υπήρχαν κάποιες τροπολογίες επί των οποίων συμφωνήσαμε, κάποιες άλλες χρειάστηκαν παραπάνω δουλειά σε ό,τι αφορά και τη διατύπωση αλλά και το περιεχόμενο. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά ακόμα. Όσο πιο πολύ συνεργαστούμε, τόσο πιο πολύ θα, τόσο πιο καλή θα είναι η συμβιβασμή που θα πετύχουμε για την επόμενη εβδομάδα. Δεν νομίζω να έχει καταφτάσει εδώ ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα copyright πνευματικών δικαιωμάτων είναι εδώ πέρα υπόλοιποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εδώ τα άτομα για το IPR. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να ενημερώσουμε ίσω οι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του συναδέλφου του για το γεγονό ότι κοιτάζουμε το θέμα αυτό πιο νωρί. Μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά σε ό,τι αφορά τη διαδικασία. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον έτσι καλά, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τη γραμματεία και νομίζω ότι πραγματικά οι συνάδελφοι θα μπορούσαν στην παρούσα φάση να σχολιάσουν να αναφέρουν ποιε είναι οι ανησυχίε του σε ό,τι αφορά τι ε, συμβαστικέ τροπολογίε. Αλλά το θέμα είναι να υποβάλουμε τα κείμενα αυτά προ τη γραμματεία για να διασφαλίσουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε επιτάπητο τι ε, συμβαστικέ προτάσει για το φάκελο αυτό. Κύριε Πάβανοβα, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προτινόμενες συμβαστικές τροπολογίες. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για πραγματική ιδιοκτησία στην ε, κοινωνία τη πληροφορία, της πληροφορίας εμπλέκονται πάρα πολλοί παράγοντες και φορείς και είναι θεωρώ ενδεικτικό το γεγονό ότι μιλάμε για τόσο πολλού ε, διαφορετικού παράγοντε και αυτό αποτυπώνεται στο κείμενο. Ελπίζω οι προτάσει να είναι αρκετά ισόρροπε. Προκειμένου να βελτιώσουμε πραγματικά το κείμενο της έκθεσης. Ήταν πολύ επικοδομητική η συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο με την κυρία Στάιλερ και τους σκιώδες εισηγητές. Σας συζητήσαμε όλες αυτές τις σημαντικές τροπολογίες και νομίζω ότι πραγματικά ήταν εξαιρετική δουλειά η εισηγητρία. Και ανυπομονώ να δω και την τελική τους εκτόχη μέχρι αύριο. Να ευχαριστήσω. Και πιστεύω γιατί, να ευχαριστήσω μάλλον τον εισηγητρία, γιατί πιστεύω ότι πολλές από τις, ε, τις ε, τροπολογίες του ΕΛΚ συμπεριληφθήσαν και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις ε, παρεμβάσεις τους. Να ευχαριστήσω την Πρόεδρο Φόρτ, την κυρία Κάλλας, την ίδια την εισηγήτρια και άλλους που κατέθεσαν κοινέ τροπολογίες. Καταρχά, πιστεύω ότι θα πρέπει να προτείνουμε μια νομοθεσία η οποία θα ενημερώσει το νόμο για τους νόμους για την πνευματική ιδιοκτησία και να την προσαρμόσει στην ψηφιακή εποχή. Ύστερα, να υπάρξει σωστή ισορροπία μεταξύ καταναλωτών, δικαιούχων και δημιουργών. Και πιστεύω ότι αυτό το πετυχαίνει ο συμβασμος ένα 1α. Τρίτο σημείο, σωστή προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, ε, καταπολεμώντα σωστά τις παραβιάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων και κάποιε άλλε τροπολογίε, πιστεύω μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά το κείμενο. Υπάρχουν 13 του κ. Ζωβάν για την μεταφορέ υπόλοιπη αξία ή 32 ή 31 και πιστεύω ότι θα πρέπει να εκτάξουμε και το θέμα της ε, φορετότητας των ε, υπηρεσιών, όπως αποτυπώνεται στην τροπολογία 41 του ΕΛΚ. Έχω και μια πρόταση την οποία θα σας την αποστείλω αργότερα για την προσθήκη μια νέα παραγράφου. Μπορώ να σας πω και την διατύπωση τώρα για την τροπολογία 79 που ήδη έχει κατατεθεί για την αναγνώριση των θεμάτων που σχετίζονται με, το πνευματικό, με την πνευματική ιδιοτησία και που σχετίζονται με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Αναγνωρίζουμε ότι αυτά είναι όλα απαραίτητα στοιχεία για τις επιχειρήσεις. Ελπίζουμε να υποστηριχθούν λοιπόν αυτές οι τροπολογίες. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνεργαστήκαν μαζί μου και προσβλέπω στις τελικές ε, τροπολογίες. Σας ευχαριστώ και καλή πτήση. And uh, Ίσως ε, να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος για να μιλήσει και για τις δύο ομάδες τροπολογιών. Η Μαρία όμως είναι η υπεύθυνη για θέματα πολιτικής ανταγωνισμού, δεν έχει καταφτάσει ακόμα. Ναι, σε λίγο. Θα έρθει ίσως, νομίζω ότι χρήσιμο θα ήταν να την ακούσουμε σε ό,τι αφορά ναι, ίσως να το κάνουμε αυτό στο τέλος. Στο τέλος της συζήτησης. Άρα συζητήσουμε και τις δύο σας ε, εκθέσεις. Από το ECR τώρα. Και εμείς δεχόμαστε πολλά από αυτά που λέει η έκθεση και ευχαριστώ την Ζητή και τους Ιωσκιώδης για την συνεργασία μας. Για μας είμαστε και υπέρ των περισσότερων συμβιβασμών, συμβιβαστικών τροπολογιών γιατί συμπεριλήφθηκε και μία δική μας τροπολογία ως προς την κατανόηση ή την ευληψία από τους καταναλωτές των κανόνων που ισχύουν για τις αδειοδοτήσεις είναι νομίζουμε πολύ σημαντικό οι καταναλωτές να γνωρίζουν τι περιορισμούς έχουν αυτές οι άδειες για να μειωθούν οι απογοητεύσεις Έχουμε όμως πρόβλημα με μία από τις συμβιβαστικές που αφορούν δημόσιες βιβλιοθήκες και την πρόσβαση online έργων που δεν έχουν κυκλοφορήσει αλέως. Δεν διαφωνούμε, αλλά ανησυχούμε με τη διατύπω, για τη διατύπωσή της που είναι κάπως ασαφής και θα μπορούσε να μειώσει τα δικαιώματα copyright ορισμένων. Εκτός αυτού είμαστε υπέρ όλων των υπολείπων και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη γενική γραμμή που παίρνει η έκθεση αυτή η γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Η εισηγήτρια. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για τις συμβιβαστικές. Νομίζω ότι οι περισσότερες από τις συμβιβαστικές είναι καλές, κάποιες μόνο χρήζουν βελτιώσεων. Η τρίτη, νομίζω ότι εδώ τα δικαιώματα των επιχειρήσεων ε, είναι ουσιαστικά κίνητρα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι αλλαγές στην πνευματική ιδιοκτησία θα πρέπει να είναι συμβατές με τις επιθυμίες των χρηστών. Αυτό θα πρέπει να φαίνεται καλύτερα στην τροπολογία 3. Στην 5 τώρα, νομίζω ότι οι εδαφικοί περιορισμοί δημιουργούν στην πολυδιάσπαση της αγοράς και γι' αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Η έκτη αναγνωρίζεται η σημασία σωστής ενημέρωσης προς τον καταναλωτή αλλά νομίζω ότι η διατύπωση μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω, διευκρινίζοντας ότι η πληροφόρηση αυτή δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε γεωγραφικές μόνο περιοχές. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ. Ρέντα. Ευχαριστώ. Είμαστε ικανοποιημένοι για τις διαπραγματεύσεις, για τις συμβιβαστικές μέχρι τώρα. Η εισηγήτρια έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά συνδυάζοντας τις διαφορετικές απόψεις. Θα συμφωνήσω με το σχόλιο του κ. Γκόργα ότι η διαφάνεια στις αδειοδοτήσεις είναι σημαντικό για να μπορεί ο χρήστης να γνωρίζει περί τίνος πρόκειται. Αλλά αυτό δεν είναι φυσικά άλοθη για την ολοκλήρωση ή στην ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Η έξι λοιπόν θα πρέπει να διευκρινιστεί καλύτερα, να πούμε ότι ναι μεν διαφάνεια είναι στόχος, αλλά θα πρέπει να βρεθούν κοινοί πραγματικά κανόνες. κάτι το οποίο θα ήταν συμβατό με τις προσδοκίες μας. Ένα θέμα το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα αφορά μία από τις τροπολογίες οι οποίες κατετέθησαν ε, για τα ηλεκτρονικά βιβλία και τον ηλεκτρονικό δανεισμό. Ε, νομίζω ότι εφόσον μπορούμε εμείς να προβλέψουμε μία ε, εξαίρεση για τα λεγόμενα e-book και ε, τον ηλεκτρονικό δανεισμό τους από τη βιβλιοθήκη. Εμείς θέλουμε τέτοιες ε, ε, συνθήκες να εφαρμόζονται και για τα ηλεκτρονικά βιβλία όπως και για τα έντυπα. Αυτό το δικαίωμα μιας επιχείρησης να αγοράζει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο και να μπορεί να το δανείζει είναι κάτι το οποίο ε, ισχύει νομίζω. Αυτό είναι εφικτό να γίνει. Υπάρχει δυνατότητα επίσης να υπάρξει και μια εξαίρεση έτσι ώστε κάποιες συμφωνίες να συνυπάρχουν μεταξύ τους, με διαφορές όμως μεταξύ τους. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει και η δυνατότητα δημιουργίας ενός ειδικού πόρταλ, μιας ειδικής ψηφιακής θύρας, ή μέσω της οποίας να μπορεί κανείς να δανείζεται ηλεκτρονικά βιβλία. Πρέπει οι βιβλιοθήκες να μπορούν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους, όπως και η αρχιοθέτηση των ηλεκτρονικών βιβλίων, έτσι ώστε να παραμένουν για την χρήση των μελλοντικών γενεών. Να περάσω τώρα στη συμβιβαστική τρία. Θα πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε ότι η εναρμόνιση σε υψηλό επίπεδο της προστασίας θα πρέπει να συνοδεύεται με τον καθορισμό των εξαιρέσεων. Εμείς δεν ζητάμε ε, κάποιες από τις ε, εξαιρέσεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα να ακυρωθούν. Νομίζω ότι όλες οι εξαιρέσεις οι οποίες υπάρχουν για τα πνευματικά δικαιώματα στα κράτη-μέλη έχουν συγκεκριμένους στόχους όπως η ελευθερία λόγου και το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Είμαι λοιπόν βέβαιη ότι θα καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία και θα έχουμε μια καλή γνωμοδότηση που θα συνεισφέρει ιδιαίτερα στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Υπάρχουν άλλα μέλη τα οποία θα ήθελαν το λόγο, όχι θα ήθελα εγώ να θέσω ορισμένα θέματα, να αναφερθώ σε πέντε τροπολογίες. Το πρώτο, για τις εξαιρέσεις. Οποιασδήποτε εξαιρέσεις υπάρξουν, θα πρέπει να είναι οικονομικά και κοινωνικά ωφέλιμες. Mm. Και θα πρέπει επίσης να είναι τεχνολογικά ουδέτερες Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να διευκρινίσουμε περισσότερο. Και για την εξαίρεση για τις βιβλιοθήκες θα έλεγα ότι κατανοώ τον λόγο για τον οποίο κάνετε αυτό το αίτημα, έχετε αυτό το αίτημα. αλλά για τα βιβλία τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα διαθέσιμα, τότε οι περιορισμοί αυτοί ίσως είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι ωφέλιμο για τις βιβλιοθήκες. Εδώ μπορούμε να διασφαλίσουμε την πολλαπλότητα του περιεχομένου που είναι ένας βασικός μας στόχος. Τώρα, ο στόχος της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ακριβώς ε, να ε, ενθαρρύνει την πολλαπλότητα του περιεχομένου και να τονώσει τη δημιουργικότητα των ε, συγγραφέων κτλ. Βλέπω εδώ την τροπολογία 29 σχετικά με την διαπραγματευτική θέση των καλλιτεχνών και δημιουργών. Φυσικά και θα πρέπει να αξιολογήσουμε σωστά τον ρόλο τους, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να διασφαλίσουμε και το ότι οι εκδότες θα πρέπει να είναι σε θέση να κερδίζουν, να υπάρχει μια προστιθέμενη αξία. Υπάρχει πάντα μια ένταση ανάμεσα στον δημιουργό και τον εκδότη, αλλά νομίζω ότι μπορούμε με την 29 να τα ρυθμίσουμε τώρα και για την, ε, την δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων. Νομίζω ότι εφόσον το περιεχόμενο το online ε, δεν θα είναι διαθέσιμο σε μία χώρα, δεν μπορεί να είναι διαθέσιμο σε άλλη χώρα. Αλλά από την άλλη κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει κάποιον να βρει το περιεχόμενο το οποίο επιθυμεί σε οποιοδήποτε άλλο μέρος αν στο δικό του δεν είναι. Δεν θα πρέπει να κάνουμε ένα αγώνα προς χαμηλότερα επίπεδα, και δεν θα πρέπει να μπορεί κανείς να επιλέγει κάποια άλλες χώρες μόνο και μόνο για λόγους τιμής. Εδώ η 14 για περισσότερη εναρμόνιση των φιλελευθέρων είναι κάτι που με ανησυχεί. Δεν ξέρω ακριβώς πού θέλουν να υπάρξει περαιτέρω εναρμόνιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της προσπάθησε να διαχωρίσει από τη μία ε, το να μην υπάρχει δυνατότητα γεωγραφικού αποκλεισμού ε, για ορισμένα περιεχόμενα, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα ιδιαίτερα περίπλοκο και ακριβό που θα περιορίζει την κυκλοφορία του περιεχομένου που μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, μίλησα πολλή ώρα, τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έφτασε, υποθέτω. Λοιπόν, μπορείτε να μας παρουσιάσετε την άποψή σας και την άποψή σας κυρίως για τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη αν ε, καθυστερήσαμε. Μα είπαν ότι προχωρούσατε γρήγορα, αλλά δεν φανταστήκαμε ότι θα πηγαίνετε και τόσο γρήγορα πια. Σου δώσω συγγνώμη. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά που είδαμε ω τώρα από την ΙΜΚΟ για το θέμα του copyright των πραγματικών δικαιωμάτων. Οι εργασίες συνεχίζονται από ό,τι καταλαβαίνω για να επιτευχθούν ε, συμβαστικές τροπολογίες και προφανώς η ΙΜΚΟ θα τονίσει τις πτυχές που σας απασχολούν πιο πολύ από όλες. Συμπεριλαμβανομένης και της ελεύθερης μετακίνησης και κυκλοφορίας των υπηρεσιών διασυνοριακή πρόσβαση σε περιεχόμενα και θα πρέπει να βρούμε μια λύση για να βελτιάσουμε τα χαρακτηριστικά αυτά και τις υπηρεσίες περιεχομένου χωρίς να εφαρμόσουμε το σύστημα πανευρωπαϊκών ε, αδειών. Αυτό νομίζω μας απασχολεί όλους και είναι κοινό μας στόχος για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και των προϊόντων, αλλά κυρίως των υπηρεσιών. Και αυτό απασχολεί όλους τους κλάδους. Είδαμε λοιπόν ε, ότι εξετάσατε διάφορες ε, σημαντικές λύσεις. Προφανώς είναι ενδιαφέρουσα η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί αυτή η συζήτηση για την έκθεση αυτή από ό,τι καταλαβαίνουμε έχει να κάνει κυρίως με τα προβλήματα εφαρμογής της ε, οδηγίας του 2001 για τις πληροφορίες. και όχι τόσο το θέμα της ανανέωσης της νομοθεσίας, το οποίο συζητιέται ακόμα μεταξύ της αρμόδιας επιτροπής και του αντιπροέδρου και δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα. Μας ζητήσατε να αναδιαμορφώσουμε το νομοθετικό πακέτο, δεν έχει όμως αυτό ακόμα αποφασιστεί. Στην παρούσα φάση λοιπόν θα πρέπει να αρκεστώ στις γενικές αρχές αν υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις από πλευρά των βουλευτών για προβλήματα που αντιμετωπίσατε σε θέματα εφαρμογής της οδηγίας του 2001, αυτό έχει απασχολήσει ιδιαίτερο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε διεξαγάγει νομικές και οικονομικές μελέτες και ευχαρίστω να απαντήσουμε σε θέματα εφαρμογής. Αλλά λοιπόν νομίζω ότι σε αυτό σε αυτά θα ήθελα να περιοριστώ στην παρούσα φάση, εκτός και να έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις και πάλι ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρησή μου. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Στάιλερ θέλει να κάνει κάποια σχόλια ίσως. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομη. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ευχαριστήσω και να πω ότι όντω δεν μπορείτε να υπολογίσετε απόλυτα τη χρονική στιγμή συζήτηση των ζητημάτων των θεμάτων στην ημερησία διάταξη, στην Επιτροπή μα. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας και τις επόμενες ημέρες θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια διατύπωση που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Να σας ευχαριστήσω όλους για την συνεργασία σας. Ήταν νομίζω πάρα πολύ εποφελή. Ελπίζω να βοηθήσουν αυτά και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Αυτές οι 550 τροπολογίες θα πρέπει να δημορφωθούν σε συμβαστικές τροπολογίες τελικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Η Πρόεδρος. Και τώρα να περάσουμε στο σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη, που είναι η γνωμοδότηση ανανεωμένη συνένεση όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανατική διεκτησία στην αστρική αγορά. Και πάλι η Κάθριν Στάιλ είναι η συγκεντρία. Εδώ είχαμε μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, την οποία κατήρτησε ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής «39 ε. ε, τροπολογίες καταθήστηκαν, έξι συμβαστικές». Να κοιτάξουμε λοιπόν τις τροπολογίες. να θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ σπουδαία ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι για τις τροπολογίες για την ε, έκθεσή μου για τις προτάσεις για το IPR. Επισκέφθηκα την υπηρεσία εναρμόνισης της ιστορικής αγοράς την εβδομάδα πριν από το Στρασβούργο. Ήταν πάρα πολύ λοιπόν ε, ωφέλιμο να δούμε τι γίνεται στο παρατηρητήριο αυτό, τι δουλειά γίνεται. Να καταλάβουμε λίγο παραπάνω τις λειτουργίες πέρα. Να καταλάβουμε μάλλον τη σημασία και το έβρος, την κλίμακα της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ευρωπαϊκή οικονομία Έχω γράψει πόσο σημαντικό είναι αυτό ό,τι αφορά την οικονομία και τι θέσει απασχόληση. Να καλέσω του συναδέλφου που δεν έχουν επισκεφτεί την υπηρεσία αυτή να το κάνουν. Και καλό θα ήταν να έρθει και κάποιο από την υπηρεσία εδώ πέρα να μα ενημερώσει. Καλό θα ήταν και οι υπόλοιποι συναδελφοί να κατανοήσουν την εργασία που γίνεται εκεί. Στις συμβαστικές τροπολογίε, έξι τον αριθμό. Και πάλι ήταν πολύ επωφελή στι συνεδρίες στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιες τροπολογίε, ξέρω ότι θα πρέπει να τι δουλέψουμε κι άλλο. Αλλά και πάλι έχουμε χρόνο μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Όπω και στο θέμα του copyright. 39 ήταν συνολικά οι τροπολογίε που κατατέθησαν. Έξι θα είναι οι συμβαστικές. Νομίζω ότι καθοδηγούν κάπως τη συζητήση μας και μια και είναι τόσο περιορισμένο περιορισμένη η εκταστή των οκτωματοτήσεων. Καλό είναι θα πρέπει να, να κοιτάξουμε τα ζητήματα αυτά, να υποστηρίξουμε αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να ακούσουμε τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις, ε, τις συμβαστικές προτάσεις, για το περιεχόμενο της γνωμοδότησης και για ενδεχόμενες ενημερώσεις ε, που μπορεί να υπάρχουν. Σας ευχαριστώ και πάλι Πρόεδρε και δυστυχώς θα πρέπει να φύγω σε λίγο για να μιλήσω, να παρευρεθώ στη συνεδρίαση για τα ψηφιακά περιεχόμενα. Θα συνεδριάσουμε και με την Ισλανδία, την Ελβετία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο στάτους και καθεστώς παρατηρητή, αλλά νομίζω πάρα πολύ ωφέλιμη αυτή η ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέει η Πρόεδρος. Um, I'll speak in the name, if you um, να μιλήσω εξ ονόματος της Κιόδους Σαμπίνας που δεν μπορούσε να προσέλθει σήμερα. Μου έστειλε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα όπου μου ζητάει να σας ευχαριστήσω ρητά για αυτή την ισορροπημένη γνωμοδότηση και την εξαιρετική συνεργασία. Για το ΕΛΚ στο σημαντικό ήταν να τονίσουμε ότι η εφαρμογή του IPR είχε στόχο να οθήσει την ανταγωνιστικότητα κλπ. Εκτός αυτού, οι παραβιάσεις έπρεπε να μεταφερθούν, να μην μεταφερθούν μάλλον, στους νέους, στην νεότερη γενιά που δεν γνωρίζουν αυτά τα πράγματα. Το ΕΛΚ εξάλλου κατέθεσε και δύο τροπολογίες ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί για αυτές χρειάζονται σαφείς δομές για την εφαρμογή αυτών των πνευματικών ή διανοητικών δικαιωμάτων και πρέπει να έχουν και πρόσθετες ρήτρε αυτές. Από την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο διαπιστώθηκε μεγάλη συνένεση στην ομάδα του Έλκαλα και μεταξύ των άλλων ομάδων και επετέχθησαν ήδη από τότε μερικές συμβιβαστικές λύσεις. Ακόμη μερικές ελάσσονες αλλαγές χρειάζονται σε αυτές, αλλά όπως είπε και η Σαμπίνα Φερχάγεν, ευελπιστούμε να βρεθεί μια λύση και για αυτές τις εκκρεμότητες. Ευχαριστώ ξανά την εισηγήτρια καθώς και τις υπόλοιπες ομάδες για τη συνεργασία. Και λέει η Σαμπίνα ξανά ότι λυπάται ιδιαίτερα που δεν είναι παρούσα. Ευχαριστούμε. Άλλη παρνόσευη, αλήπη. Αν θα την αντικαταστήσεις είπες. Ο Ντάλτον, ο Ντάλτον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως και για το προηγούμενο θέμα, είχαμε πάλι πολύ καλή συνεργασία μεταξύ σκιωδών. Για μας η εφαρμογή, των, η άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής διοκτησίας είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για τις δημιουργικές βιομηχανίες αλλά και για άλλους τομείς. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Υπάρχουν διαφορές όμως μεταξύ ε, των παρατυπιών που σημειώνονται online και offline και αλλιώς τα βλέπει και το κοινό. Στις offline παρατυπίες φαίνεται πολύ περισσότερο πιο γρήγορα ότι πρόκειται για παρατυπία από ό,τι στις online. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε σφαιρικά και να δούμε τι επηρεάζει το θέμα αυτό των παρατυπιών. Μπορεί κάποιος να θέλει πρόσβαση σε κάποιο περιεχόμενο χωρίς να παραβιάζει τα δικαιώματα και να θεωρείται τεχνικός ως παραβίας. Στο σχέδιο δράσης της Κομισιόν και τώρα και στους συμβιβαστικές ακολουθήσαμε την γραμμή follow the money να δούμε δηλαδή ποιοι εκμεταλλεύονται, ποιοι κερδίζουν από τις παρατυπίες. Από τις περισσότερες συμβιβαστικές είμαστε ικανοποιημένοι, έχουμε όμως και μερικές αμφιβολίες, κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο η συμβιβαστική για το back είναι διατυπωμένη. Εμείς θα προτιμούσαμε μία, να δούμε πρώτα ποια είναι τα στοιχεία και μετά να καταλήξουμε σε συμπέρασμα. Εκτός αυτού όμως είμαστε γενικά ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η Ντίτα Σάντσοβα. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγητή. Και εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με ό,τι έχει γίνει για αυτήν την με αυτό το θέμα. Και μετά τη τελευταία συνάντηση των σκιωδών νομίζω ότι θα τα δεχτούμε όλα. Γενικά σχεδόν όλες οι τροπολογίες είναι θετικές αλλά δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε όλες, τελείως όλες. Μία ας πούμε για τη σημάνσεις, η 34, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Γιατί εδώ μιλάμε για παρατυπίες στην άσκηση των πνευματικών δικαιωμάτων ενώ εκείνη μιλάει για καθαρή παρανομία και αντιγραφή. Δεν νομίζω ότι η ιδέα των ψηφιακών ετικετών ή badges βοηθάει. Κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα ούτε θα υπάρξει στην ψηφοφορία. Ζούλια γιατί δεν έχουμε κανέναν από την Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμβιβαστική λύση, αποδοχή της συμβιβαστικής λύσης οι απόψεις μας έγιναν δεκτές, αντικατοπτρίζονται στις προτάσεις της εισηγήτριας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτά τα οποία είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι για το τι εννοούμε ε, με τη συμφωνία αυτή. Η πνευματική διοκτησία είναι ένα μικρό πνεύμα, μια ευρύτερη, ένα μικρό τμήμα μια ευρύτερη προσπάθεια. Ε, έχουμε πολλά να κάνουμε και με άλλες μορφές παραβίασης ή προσπάθειας παραβίασης ε, ε, των κανόνων. Πρέπει να γίνουν πολλά και στον τομέα της προστασίας των διπλωμάτων τα κτλ. Τώρα για τις συμβιβαστικές έχουμε ένα θέμα μόνο με την τρία το οποίο συζητήσαμε αλλά δεν έχουμε καταλήξει ακόμα για τη συμπερίληψη ε, ενός συστήματος προειδοποίησης των καταναλωτών. Ε, για μας δεν είναι ξεκάθαρο αν τέτοιο σύστημα, αν ένα τέτοιο σύστημα ε, αφορά ένα σύστημα προειδοποιήσεων σαν παράδειγμα σε τρεις φάσεις που μπορεί να οδηγήσουν και στο να σταματήσει η σύνδεση με το διαδίκτυο στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει ε, μια διόρθωση της συμπεριφοράς κάποιου χρήστη. Λοιπόν, πέραν αυτού όμως ε, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις συμβιβαστικές τροπολογίες ως έχουν. Ένα σημείο να προσθέσω εδώ που συζητήσαμε στους σκιώδεις και είναι ωφέλιμο για όλους. Τέθηκε μια ερώτηση για την 30 από ορισμένους συναδέλφους για την ανάγκη που υπάρχει για εντοπίσιμες πληροφορίες ε, για αυτόν ο οποίος ε, είναι ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένη ψηφιακή διεύθυνση. Αν υπάρχει ένα βιβλίο ή ένα προϊόν, υπάρχει ένα trademark ε, με μια ευρεσιτεχνία, μια κάτι υπάρχει. Πολλές φορές όμως για το ψηφιακό περιεχόμενο κάτι τέτοιο δεν είναι δεδομένο. Αν υπάρχει μία εικόνα βέβαια ε, στο διαδίκτυο δίδεται μία πληροφορία για την εικόνα αυτή. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την δυνατότητα εντοπισμού συγκεκρισμένων ε, στοιχείων και μέσω της συμπερίληψης των λεγόμενων ε, μεταδεδομένων, κάτι το οποίο θα διευκολύνει κατά πολύ την έβρεση των περαιτέρω στοιχείων. Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε μέσω μιας προφορικής τροπολογίας. Μιλάμε για μεταδεδομένα και όχι για τη δημιουργία σώνει και καλά μια τεράστιας βάσης δεδομένων. Έχουμε και ένα επιπλέον εισηγητή από το FDD αλλά δεν είναι παρόν. Λοιπόν, θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σύντομα. Δεν έχουμε δει τις συμβιβαστικές ακόμα, αλλά ακούσαμε αυτά τα οποία είπαν οι διάφοροι κοινοβουλευτικοί. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κάποια συνένεση Ε, ελπίζω να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση. Δύο στοιχεία τα οποία μπορεί ίσως να βοηθήσουν. Ε, σχετικά με την 34 και τις ετικέτες, την επισήμανση. Ε, οι κατάλογοι μπορεί να είναι ένα πρόβλημα βέβαια και το να συμπεριληφθούν αυτά τα στοιχεία αλλά αυτό δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση που μπορεί να υπάρξει. Πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες και σε σχέση με το IP Μερικά από τα δεδομένα αυτά φαίνονται βέβαια πάρα πολύ χρήσιμα αλλά μπορεί να δημιουργούν προβλήματα. Δεν ξέρω τι υπόθηκε ακριβώς προηγουμένως για το ότι αυτό το πρόγραμμα δράσης ε, καλύπτει όλες τις παραβιάσεις IP ε, και σε εμπορικό επίπεδο. Πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ακριβώς οι εμπορικές κλίμακες και να προσπαθήσουμε να τις αποφύγουμε. θα πρέπει να υπάρχουν όπως είπαμε και ε, διαιτητικές ή ε, ενδιάμεσες υπηρεσίες που θα επιτρέπουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναζητούν στοιχεία και να προσπαθούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Σας ευχαριστώ ε, που μας υπενθυμίσατε ότι δεν πρόκειται για θέματα αμοιβής μόνο, αλλά και για θέματα ασφάλειας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και δική μου επίσκεψη στην υπηρεσία και καλό θα είναι να, να μην υπάρχει άλλη και να υπάρχει μια διαδικασία εντοπισμού των παραβιάσεων. Ίσως λοιπόν τέτοιου είδους ε, οργανώσεις, υπηρεσίες θα πρέπει να καλούμε στην Επιτροπή μας. Η ε, κάθε τώρα έχει το λόγο για να σχολιάσει εν συντομία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε για το θέμα της πρόσβασης. Ε, τα πέρα λοιπόν τα τα παραβίασης ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Καλό είναι λοιπόν να προωθήσουμε τι έξι αυτέ συμβαστικές τροπολογίε. Ευχαριστώ και πάλι του συναδέλφου για τη συνεργασία για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι όταν περνάμε σε θέματα ουσία, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό, όχι μόνο για την εκάστοτε εκλογική περιφέρεια, αλλά για όλη την ευρωπαϊκή κοινότητα. Νομίζω ότι το εύρο και η κλίμακα του θέματο αυτού είναι κάτι το Πρωτοφανέ. Είναι καλό λοιπόν ε, που υπάρχουν και προτείνονται αυτά τα μέτρα εφαρμογή και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να βρούμε ποιοι βρίσκονται στον πυρήνα των παρεμβιάσεων αυτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, προσβλέπω στα σχόλιά σας και στις ψηφοφορίες την επόμενη εβδομάδα. Και έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή συνεδρίαση και ξεκινάμε πάλι αύριο στις 9 για να συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης για το TTIP. Είμαι βέβαιη ούτε, αυτό θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα.